Αγαπητοί συνάδελφοι, καλημέρα σας. Καλωσορίζω τον Χερούν Ντέιζελμπλουμ. Όπως ξέρετε, είναι σήμερα στην Επιτροπή μας, όχι υπό την ιδιότητα του Προέδρου του Eurogroup, αλλά ως Πρόεδρος του ΕΚΟΦΗΝ αυτό το εξάμεινο. Και έχουμε την ακρόασή μας, όπου θα μας παρουσιάσει τα αποτελέσματα της Ολλανδικής Προεδρίας για θέματα αρμοδιότητας ε, της Επιτροπής μας. Από πλευράς μας λοιπόν, ευχαριστώ τον κύριο Ντάισελμπλουμ για το πνεύμα συνεργασίας που επεδείχθη κατά την Προεδρία της Ολλανδίας. Ε, συνεχίσαμε να εργαζόμεθα για σημαντικά θέματα όπως η Ένωση Κεφαλαγορών Έντις, ΑΙΟΠΑ, με θετικά αποτελέσματα να αναμένονται τους επόμενους μήνες ή και τις επόμενες μέρες. Αύριο έχουμε τη σημαντική και ελπίζω τελική συνάντηση τριμερούς διαλόγου για το ΑΙΟΠΑ. Για τον τομέα της προλογίας χαιρετίζουμε τη φιλόδοξη προσέγγιση της Ολλανδικής Προεδρίας. Θέλησε να προωθήσει τα θέματα φορολογίας ως Κοινοβούλιο. Θα θέλαμε να ληφθεί σοβαρότερα υπόψη από το Συμβούλιο ε, ο ρόλος μας μέσω της ε, διαβούλευσης και για το πακέτο κατά της φόρο αποφυγής έχουμε ένα κείμενο ρωμαλαίο και φιλόδοξο που ελπίζω να ληφθεί υπόψη και οπωσδήποτε θα καθορίσει ε, αυτά που θα μας απασχολήσουν στα επόμενα βήματα. Σύμφωνα με τις συνήθεις διαδικασίες θα έχουμε μία εισαγωγική δήλωση 10 λεπτών από τον κύριο Ντάισελμπλουμ και μετά θα έχουμε τη συνήθη διαδικασία ερωταπαντήσεων. Χαιρούν, έχεις το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Αγαπητά μέλη, με μεγάλη χαρά σας συναντώ πάλι εσάς στην Επιτροπή σας, την ΕΚΟΝ και με μεγάλη χαρά θα ανταλλάξω απόψεις μαζί σας. Θα υπογραμμίσω την πρόοδο την οποία έχουμε σημειώσει στα πλαίσια της Προεδρίας του ΕΚΟΦΗΝ. Είναι αρκετά νωρίς βέβαια, θα έπρεπε να γίνει αυτή η συνάντηση αργότερα γιατί την Παρασκευή έχουμε κι άλλο εκοφήν, έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας και έχουμε φιλόδοξο πρόγραμμα το οποίο σας είχαμε παρουσιάσει στην αρχή της Ολλανδικής Προεδρίας. Η προσπάθεια η οποία έχει γίνει τους τελευταίους μήνες έχει γίνει σε ένα κλίμα, θα έλεγα, οικονομικής ανάκαμψης, το οποίο συνεχίζεται σε χαμηλούς ρυθμούς, πάντως συνεχίζεται. Και αν δείτε ακριβώς αυτή την οικονομική ανάκαμψη, θα καταλάβετε ότι έχουμε ανάγκη από μια μορφή ανάπτυξης βιώσιμη εκ των έσω περισσότερο, ιδιαίτερα βλέποντας τα εξωτερικά προβλήματα, όπως την ιδιαίτερα χαλαρή νομισματική πολιτική, όπως επίσης και τις χαμηλές τιμές του πετρελαίου. Πρέπει να ενισχύσουμε την ε, οικονομία μας και την οικονομία της Ευρωζώνης ειδικότερα. Αυτό υπογραμμίζει τη σημασία του συντονισμού των ευρωπαϊκών πολιτικών. Πρέπει να ενισχύσουμε τις διαφορετικές μεταρρυθμίσεις, τις επενδύσεις, να έχουμε αποτελεσματικές δημοσιονομικές πολιτικές και ε, ε, υγιείς τομεακές πολιτικές έτσι να μειώσουμε την απαράδεκτα υψηλή ανεργία σε, άλλες, σε πολλές χώρες και άλλες απαράδεκτες μορφές κληρονομιάς, θα έλεγα, της οικονομικής κρίσης. Πιο συγκεκριμένα, εμείς έχουμε επεξεργαστεί κάποιες νομοθετικές προτάσεις. Να κάνω καταρχάς κάποιες παρατηρήσεις όμως για την προσπάθεια την οποία κάνουμε στα πλαίσια της έκθεσης των πέντε Προέδρων. Καταρχάς, ολοκλήρωση της ε, Τραπεζικής Ένωσης. Αυτό είναι ένα από τα θέματα που θα συζητήσουμε την ε, Παρασκευή στο ΕΚΟΦΗΝ. Έχουμε πετύχει αρκετά. Ο πρώτος πυλώνας και ο ενιαίος μηχανισμός επίβλεψης, το SSM, ήδη ε, είναι κομβικός παίκτης ο δεύτερος πυλώνας για την αντιμετώπιση των προβληματικών τραπεζών θα αρχίσει να εφαρμόζεται σύντομα και ήδη έχουν υπάρξει οι πρώτες καταβολές όπως επίσης έχουμε προχωρήσει και στα πλαίσια της Ευρωπα... του Ευρωπαϊκού Προγράμματος για την Εγγύηση των Καταθέσεων. Περισσότερα πρέπει να γίνουν στο μέλλον ιδιαίτερα σχετικά με τον τρίτο πυλώνα. Έχει ξεκινήσει μια ομάδα εργασίας της συζητήσεις τον Ιανουάριο επί τη βάση των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Ευρωπαϊκό Σχέδιο για το Πρόγραμμα Εγγυήσεων, τη μείωση των κινδύνων και την ισότιμη και δίκαιη ανταγωνιστικότητα στον πιστοτικό τομέα. Υπάρχουν αρκετά περίπλοκα θέματα Έχουμε οργανώσει τη δουλειά μας έτσι ώστε η μείωση των κινδύνων και η κατανομή των κινδύνων να είναι δύο πρωτοβουλίες που ακολουθούν παράλληλη πορεία. Τους τελευταίους μήνες η ανταλλαγή απόψεων μας επέτρεψε να κατανοήσουμε καλύτερα τις διάφορες ευαισθησίες και τα τεχνικά θέματα και διαφοροποίησεις γύρω από τα θέματα αυτά. Στόχος μας είναι να υπάρξει μια συμφωνία για το πώς θα συνεχίσουμε από εδώ και πέρα τα επόμενα χρόνια ήδη από την επόμενη Παρασκευή στη συνάντηση του ΕΚΟΦΗΝ. Αυτό θα υπογραμμίσει λοιπόν τη δουλειά που θα κάνουμε και στα πλαίσια της κατανομής κινδύνου και στα πλαίσια της μείωσης του κινδύνου και πρέπει να βρεθεί μια σωστή ισορροπία ανάμεσα στα διαφορετικά συμφέροντα και στις διάφορες χώρες. Τώρα για την Τραπεζική Ένωση είναι ένα θέμα που περιλαμβάνεται στην έκθεση των πέντε πρόεδρων. Από την άλλη έχουμε και την αγορά κεφαλαίων. Και εδώ περιμένω από το ΕΚΟΦΗΝ της Παρασκευής να επιβεβαιώσει τη συμφωνία για τις θέσεις του Συμβουλίου, για τον κανονισμό για τα ενημερωτικά δελτία. Ελπίζω λοιπόν να ξεκινήσουμε τις ε, τριμερείς διαπραγματεύσεις με το Κοινοβούλιο σύντομα. Προσπαθούμε επίσης να περάσουμε και στην τελική φάση των διαπραγματεύσεων ανάμεσα στους συνομοθέτες για την πρόταση για τα όργανα για επαγγελματικές συντάξεις, η ΑΙΟΠΑ η γνωστή. Το έχετε ήδη αναφέρει και εσείς Πρόεδρε και ελπίζουμε να γίνει σύντομα αύριο. Μάλιστα προβλέπεται η τελευταία συνάντηση του τριγωνικού διαλόγου. Ελπίζω να κλείσει εκεί η διαδικασία. Υπάρχει επίσης και το πακέτο τιτλοποίησης, είναι πολύ σημαντικό θέμα της ενιαίας αγοράς κεφαλαίων, θα ωφελήσει πολύ την πραγματική οικονομία. Το Συμβούλιο έχει ήδη συμφωνήσει για μια διαπραγματευτική εντολή, ήδη από πέρυσι, και ελπίζω το Κοινοβούλιο σύντομα να ολοκληρώσει την εξέταση των προσπαθειών του για να ξεκινήσουν οι τριγωνικοί διάλογοι. Να σταθώ τώρα σε κάποια μη χρηματοδοτικά, χρηματοοικονομικά συγγνώμη, θέματα σε σχέση με την ολοκλήρωση της νομισματικής ένωσης. Υπάρχουν οι εθνικοί πίνακες ανταγωνιστικότητας, όπως γνωρίζετε, αυτό είναι κάτι στο οποίο εμείς εμένουμε σαν Προεδρία με βάση τη θετική εμπειρία που έχουμε στη χώρα μας, στην Ολλανδία. Ε, με χαρά ε, λέγω ότι προβλέπουμε να καταλήξουμε σε μια συμφωνία για την πρώτη σύσταση στο ΕΚΟΦΗΝ την προηγούμενη, αυτή την εβδομάδα. Εμείς προσπαθούμε να συγκεντρώσουμε την προσοχή μας στις εξελίξεις στον τομέα της παραγωγικότητας και όχι μόνο της ανταγωνιστικότητας σε επίπεδο κόστους. Η σύσταση λαμβάνει επίσης υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά των διαδικασιών καθορισμού των μισθών σε εθνικό επίπεδο, όπως επίσης και τους ε, προερχόμενους από αυτά νομικούς περιορισμούς. Οι πίνακες ανταγωνιστικότητας δεν είναι τα μόνα μέσα πάνω στα οποία θα έχουμε κάνει σημαντική πρόοδο για σωστές διαφορετικέ πολιτικές. Το Συμβούλιο έχει συμφωνήσει και για τη διαπραγματευτική εντολή και για ένα διαφθρωμένο μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα στήριξη το SRSP, επί τη βάση τη εμπειρία που πήραμε από ορισμένε χώρε τα προηγούμενα χρόνια. Θέλουμε να διευρύνουμε την δυνατότητα τεχνικής βοήθειας προς τα κράτη-μέλη τα επόμενα χρόνια, επαναλαμβάνω, για να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητα και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Περιμένουμε και τη δική σας θέση. Θα επιβεβαιώσουμε επίσης και μια γενική θέση του Συμβουλίου ε, για τα ταμεία των χρηματαγορών αύριο. Το Κοινοβούλιο εδώ είναι πιο μπροστά από μας και μας περιμένετε σε αυτή την περίπτωση. Ελπίζω να τα επιβεβαιώσουμε αυτά αύριο και να ξεκινήσουμε μεταξύ μας συζητήσεις. So. Και για τα φυλάδια ελπίζω να καταλήξουμε σύντομα. Τώρα τι άλλα θέματα έχουμε. Μετά από ετοιμά μας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει ένα πρόγραμμα δράσης για την χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, για το βρώμικο χρήμα. Αυτά θα τα συζητήσουμε την Παρασκευή. Έχει υπάρξει πάντως σημαντική πρόοδος, ιδιαίτερα σε σχέση με την εφαρμογή των υπαρχουσών νομικών ρυθμίσεων. Τέλος, στο θέμα της φορολογίας. Το προηγούμενο μήνα πετύχαμε λοιπόν και προωθήσαμε μία από τις βασικές προτεραιότητες, την αναθεωρημένη οδηγία για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών, το λεγόμενο DAC4. Είμαι πεπισμένος ότι αργότερα αυτή την εβδομάδα θα καταλήξουμε σε μία συμφωνία και για την οδηγία ATAD για την φοροαποφυγή. Σχετικά με το μη νομοθετικό κομμάτι του πακέτου για την φοροαποφυγή, τον προηγούμενο μήνα το ΕΚΟΦΗΝ θέτησε τα συμπεράσματα του Συμβουλίου ζητώντας να υπάρξει μια ευρωπαϊκή μαύρη λίστα μη συνεργαζόμενων ε, τρίτων χωρών, δικαιοδοσιών τρίτων χωρών. Είναι κάτι το οποίο ε, είναι όλο και πιο σημαντικό για τη δουλειά μας. Έχουμε κάνει επίσης σημαντική πρόοδο και στον τομέα του ΦΠΑ. Μια συμφωνία επί της ουσίας έχει υπάρξει σε σχέση για τα λεγόμενα vouchers που έγινε αντικείμενο διαπραγμάτευση στο Συμβούλιο ήδη από το 2012. Έχουμε πάρει λοιπόν κάποιες πρώτες αποφάσεις για το πρόγραμμα δράσης για το ΦΠΑ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ε, έχουμε συζητήσει τα κατεπήγοντα μέτρα για την καταπολέμηση της, απάσης, της απάτης των απατών γενικότερα στα πλαίσια του ΦΠΑ. Δεν θα ε, μακρηγορήσω. Έχουμε δουλέψει σκληρά πάντως μέχρι τώρα Ελπίζω να μπορέσουμε στο μέλλον να δουλέψουμε ακόμα πιο σκληρά και να συνεχίσει τη δουλειά και η επόμενη Προεδρία και να συνεχίσει και τις διαπραγματεύσεις που έχουν ξεκινήσει. Ο Πρόεδρος Γκουαλτιέρη, σας ευχαριστώ πολύ. Όντως έχετε δουλέψει σκληρά για έναν αριθμό θεμάτων. Ακόμα δεν έχω λάβει την τελική μορφή. Για το Ταμείο Κεφαλαίου Αγορών, χρήματα αγορών, διευρύνεται επίσης το πεδίο εφαρμογής για τα Συμβούλια Ανταγωνιστικότητας και αναμένουμε βεβαίως τα συμπεράσματά σας για την Τραπεζική Ένωση στο τέλος της εβδομάδας. Σας ευχαριστώ πολύ. Μπορούμε να αρχίσουμε τώρα με, την, με τον κατάλογο των εγγεγραμμένων. Πρώτη κυρία Ντέλαγκε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ίσως είναι ο καλβινιστικός μου χαρακτήρας. Μου αρέσει όμως, αρέσει το Λαϊκό Κόμμα να ακούω τον ε, ε, κύριο Ντάισερ που να λέει ότι δουλέψαμε θα δουλέψουμε ακόμα περισσότερο. Είπατε και εσείς κύριε Πρόεδρε. Ήταν φιλόδοξη η Ολλανδική Προεδρία και στον τομέα σας. Ελπίζουμε να σας ξαναδούμε πολλές φορές ε, στον ρόλο σας ως Προέδρου της Ευρωομάδας. Ένα ε, θέμα που με απασχολεί και κάτι είπατε σχετικά σε δημοσιογράφους, σχετικά δηλαδή με την αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ό,τι αφορά την εφαρμογή του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Έχετε έλθει σε επαφή ειδικά για το θέμα αυτό με την Κομισιόν και ποια ήταν η αντίδρασή τους και γιατί έχει τόση σημασία για σας. Θα θέλαμε να το ξέρουμε, διότι συμφωνούμε με την ανάλυση ότι είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι η βάση την οποία έχουμε θα διατηρηθεί. Σε ό,τι αφορά το επικείμενο ΕΚΟΦΗΝ... και βέβαια το ΕΝΤΙΣ... αύριο θα έχουμε το δικό μας έγγραφο εργασίας έτοιμο από τη δική μας πλευρά. Αποτέλεσε πρόκληση, όπως και για σας, να συμπεριλάβουμε τις διάφορες θέσεις και βεβαίως και όλα τα διασυνδεόμενα θέματα, κάποια περισσότερο, κάποια λιγότερο, σίγουρα. Είπατε ότι αναμένεται να υπάρχει συμφωνία την Παρασκευή σε ό,τι αφορά την περαιτέρω πορεία για τα επόμενα χρόνια αυτό ηχεί κάπως ως οδικός χάρτης. Δηλαδή ότι οι δύο τροχές, μείωση του κινδύνου και ε, κατανομή του κινδύνου θα κινηθούν παράλληλα. Μπορείτε να εξηγήσετε λίγο περισσότερο. Είπατε επίσης ότι η BRRD και η CSD δεν εφαρμόζονται, νομίζω από τρεις χώρες μέλη. Μπορείτε να πείτε πότε αναμένετε να εφαρμοστούν. Για να προχωρήσουμε με το έντις εμείς πρέπει να έχουμε τα βασικά στοιχεία στη θέση τους. Για το θέμα των δύο ατζέντα που πάνε χέρι-χέρι, πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι το risk reduction, αν δεν προχωρήσει αρκετά γρήγορα, διότι δεν μπορούμε να προχωρήσουμε με το έντις καθόλου. Εγώ θα ήθελα να προχωρήσουμε με το έντις. Πώς μπορούμε λοιπόν να εξασφαλίσουμε ότι θα, υπάρχει, θα υπάρχουν ε, τα αναγκαία στοιχεία ώστε να διασφαλιστεί η πορεία του σειρμού. Και ε, να μπορούμε να παρακολουθούμε και τις διεθνείς εξέλιξεις, διακόπτη ο πρόεδρος Κουαλτιέρη. Μάλιστα, τελείωσα. Ευχαριστώ, λέει ο κύριος Στάσελμπλουμ, για το πρώτο θέμα, αξιοπιστία δηλαδή, του συμφώνου και ρόλος της Επιτροπής. Θα είμαι ειλικρινής. Ανησυχώ πολύ. Όταν έχουμε συμφωνίες μεταξύ μας, είναι σημαντικό βέβαια όλοι μας να συμμορφωνόμαστε. Βεβαίως υπάρχει κάποια ευκαμψία, ευελιξία. Έχει καλώς. Εγώ μάλιστα είπα ναι, να υπάρχει ευκαμψία σε ό,τι αφορά τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Σύμφωνοι. Εδώ όμως ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καθίσταται κρίσιμος. Εάν οι χώρες μέλη θεωρούν ότι οι αποφάσεις της Κομισιόν είναι δυσνόητες και δύσκολο να προβλεφθούν και δεν είναι αντικειμενικές ή διακρίνουν μεταξύ μικρών χωρών μελών και μεγάλων χωρών μελών. Αυτό αποτελεί πηγή μεγάλης ανησυχίας. Και το νιώθω αυτό και στις συνεδριάσεις του Eurogroup ότι και οι υπουργοί ανησυχούν. Νομίζω λοιπόν ότι η Κομισιόν οφείλει να κατανοήσει ότι έχει το σύμφωνο στα χέρια της. Αυτή είναι οι θεματοφύλακες του συμφώνου, της Επιτροπής δηλαδή. Υπάρχει εντύπωση ότι υπάρχει διακριτική μεταχείριση ανάμεσα σε διάφορε χώρε μέλη και ανάλογα σε, με διάφορε καταστάσει. τότε ε, θα είναι δύσκολο να συμμορφώνονται όλοι με τα όσα έχουμε συμφωνήσει. Ωραία. Το έχω πει αυτό, το είπα και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ευθέω στου επιτρόπου γνωρίζουν την ανησυχία μου αυτή. Συμφωνούν ότι ο ρόλος τους είναι σημαντικός και ότι πρέπει να είναι αντικειμενικοί. Δηλαδή γενικά συμφωνούμε. Κάθε φορά όμως που έχω την ανησυχία αυτή θα την εκφράζω. Διότι και ο Μάριο Ντράγκη αποκαλεί το σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης την άγκυρα της σταθερότητας. Χρειάζεται λοιπόν εμπιστοσύνη όχι μόνο προς τα έξω αλλά και μεταξύ μας, μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης. Άρα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη. Για το έντις πράγματι αυτό για το οποίο μιλούμε είναι ένας οδικός χάρτης. Έτσι το αποκαλέσαμε και εμείς. Μέχρι το 2024, τον είπε 14 στην αρχή ο Μέχρι το 2024 λοιπόν θα έχει ολοκληρωθεί. Η Τραπεζική Ένωση είπαμε ότι θα μπει και ένα backstop. Θεωρώ επίσης ότι τμήμα θα πρέπει να αποτελέσει και το πρόγραμμα εγγύσεις καταθέσεων. Αυτό βέβαια ακόμα θα το διαπραγματευτούμε και θα συμφωνήσουμε. Πώς θα φτάσουμε τώρα στο 2024. Εκεί χρειάζεται πολύ δουλειά ακόμα. Και γι' αυτό η δική μας προσέγγιση είναι ότι πρέπει να είναι ισορροπημένη η προσπάθεια, πρέπει να κινηθούν και οι δύο πλευρές της ατζέντα, να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε κάποιες κληρονομιές που έχουμε στις τράπεζες ακόμα, να μειωθούν οι κίνδυνοι και ταυτόχρονα να ενσωματώνουμε όλο και περισσότερο τον ε, χρηματοπιστωτικό κανονισμό και τα ε, διάφορα προγράμματα ή συστήματα ασφαλίσεων. Εξακολουθούμε να το επεξεργαζόμαστε το θέμα αυτό. Θεωρώ πάντως ότι μπορούμε να πετύχουμε. Και τότε θα έχουμε τον οδικό χάρτη για τα επόμενα χρόνια. Όμως έχουμε πολλή δουλειά ακόμη. Οφείλετε να το αντιληφθείτε. Το αντιλαμβάνεστε νομίζω πολύ καλά πόσο δύσκολες δηλαδή είναι οι συνομιλίες αυτές, πόσο διαφορετικά είναι τα συμφέροντα, που είναι πολύ σημαντικά. Θα συνδέσουμε λοιπόν τα δύο τμήματα αυτά της ατζέντα, ώστε να επιτελέσουμε πρόοδο και από τις δύο πλευρές, με στόχο πάντοτε αυτή τη σημαντική χρονολογία του 2024. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Ντάιζελμπλουμ, Αναφέραστε στο λόγο της Κομισιόν για την εφαρμογή του Συμφώνου Σταθερότητας. Μήπως υπονοείτε με τον τρόπο που κάνετε αυτές τις αναφορές ότι η Κομισιόν είχε αυθαίρετο τρόπο εφήρμοσε τους κανόνες αυθαίρετα. Έτσι θα δημιουργηθεί το κλίμα εμπιστοσύνης. Πρέπει να υπάρχει σαφήνεια. Υπονοείται ότι δεν εφάρμοσε σωστά η Κομισιόν τους κανόνες. Δεύτερη ερώτηση. Αναφερθήκατε στα, συμβούλια, στα Εθνικά Συμβούλια Ανταγωνιστικότητας που συζητάτε στο Συμβούλιο. Θεωρείτε ότι είναι φυσιολογικό ότι δεν ε, συμμετέχει καθόλου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στη συζήτηση που θα είναι ένας από τους σημαντικούς πυλώνες της λειτουργίας της ε, οικονομικής διακυβέρνησης. Τέλος, για το έντις εγγύηση καταθέσεων. Απαντήσατε στην Ντελάνια ήδη, αλλά χθε ακούσαμε την Ντανιέλ Νουρή, η οποία μας είπε πόσο σημαντικό είναι αυτό το νομοθέτημα, ούτως ώστε να διασφαλίσουμε τη σταθερότητα των ε, χρηματοπιστωτικών αγορών και ε, μια σωστή ισορροπία. Δεν θεωρείτε ότι το χρονοδιάγραμμα που μας παρουσιάζεται είναι κάπως ε, αργό, ούτω ώστε να επανέλθει για την Τραπεζική Ένωση αυτή η εμπιστοσύνη, μάλλον να δημιουργηθεί. Γιατί αν δεν ολοκληρωθεί η Τραπεζική Ένωση ε, δεν θα είναι σταθερό το σύνολο και τίθενται εν κινδύνο αυτά που έχετε κάνει για τους δύο πρώτους πυλώνες. Ο κύριος Ντάζελμπλουμ. Ευχαριστώ κύριε Μπερέζ. Εφαρμόζει σωστά η Κομισιόν τους κανόνες. Ε, τότε δεν θα έπρεπε να το πει το ΕΚΟΦΗΝ. Έτσι δεν λειτουργεί το σύστημα. Έχουν υπάρξει κάποιες ανησυχίες για κάποιες πρόσφατες ε, αποφάσεις για τα CSR, για τις ε, συστάσεις αναχώρα. Τίθενται λοιπόν θέματα γι' αυτό αν εφαρμόζονται σωστά οι κανόνες. Ε. Το συζητήσαμε στο ΕΚΟΦΗΝ, παρουσία της Κομισιόν, για το, γιατί αντιμετωπίζεται διαφορετικά η Γαλλία. Δεν ακούμε την κυρία Μπερέζ έκανε ένα σχόλιο ο πρόεδρος, συνεχίζει ο κύριος Ντάζεμπλουμ, ότι η Γαλλία φαίνεται ε, αξίζει διαφορετικής ε, αντιμετώπισης γιατί είναι η Γαλλία. Ε, κάναμε προσπάθεια και εγώ και άλλα κράτη-μέλη να καταλάβουμε τι σημαίνει ένα τέτοιο σχόλιο και αυτό σχετίζεται με ορισμένες ανησυχίες που έχουν κάποια κράτη-μέλη, κυρίω τα μικρά, ότι τα μεγάλα κράτη-μέλη αντιμετωπίζονται διαφορετικά. Αυτό δεν είναι καλό, γιατί δεν δημιουργεί σχέση εμπιστοσύνη μεταξύ μα. Αυτό που λέω είναι ότι η Κομισιόν πρέπει να είναι πολύ προσεκτική. Είναι θεματοφύλαξη των κανόνων, είναι θεματοφύλαξη του συμφώνου, που είναι πολύ βασικό να εφαρμόζεται το σύμφωνο για να υπάρχει σωστή συνεργασία και εμπιστοσύνη για το ρόλο του Κοινοβουλίου για τα Συμβούλια ανταγωνιστικότητα. Θα έπρεπε να το έχω πιο πολύ υπόψη μου. Αλλά, κοιτάξτε, το Κοινοβούλιο δεν έχει ρόλο για αυτή την πρόταση. Δυστυχώς. Δυστυχώς. Ναι. Δεν καταλαβαίνω γιατί το Κοινοβούλιο να μην έχει ρόλο για το θέμα αυτό. Ίσως υπάρχει κάποιος νομικός λόγος τον οποίο δεν κατανοώ. Θα το κοιτάξουμε για την Τραπεζική Ένωση. Ότι προχωράμε αργά. Ίσως έχετε δίκιο αλλά ήταν σκόπιμο να υπάρξει επαρκής χρόνος για να έχει επαρκής πόρους το Ταμείο Εξυγίανσης γιατί δεν ήταν εύκολο να πάρουμε λεφτά από τις τράπεζες για να χρηματοδοτηθεί αυτό το Ταμείο και το ίδιο ισχύει και για το πρόγραμμα εγγύησης των καταθέσεων. Υπάρχουν και πολλά θέματα του παρελθόντος για τις τράπεζες που πρέπει να τα αντιμετωπίσουν. Αν θέλουμε να επιταχυνθεί η διαδικασία για να αντιμετωπίσουμε τα μη ε, εξυπηρετούμενα δάνεια ή την υψηλή συγκέντρωση δημοσίου χρέους. Δεν νομίζω ότι θα τα σκόπιμο να επιταχύνουμε. Τα θέματα αυτά του παρελθόντος θέλουν το χρόνο τους για να αντιμετωπιστούν. Και αυτό το χρόνο μπορούμε να, τα αξιοποιήσουμε, να τον αξιοποιήσουμε για να δημιουργήσουμε και αυτόν τον τελευταίο πυλώνα της Τραπεζικής Ένωσης. Πρόεδρος. Ευχαριστώ. Μπέρντ Λούκε. Εγώ θα μιλήσω γερμανικά. Κύριε Ντάισελμπλουμ, στην Γερμανία και εμείς εκτιμούμε και όχι μόνο οι καλβινιστές τη σκληρή δουλειά. Την εκτιμούμε λοιπόν όλοι. Βέβαια, η σκληρή δουλειά να γίνεται στη σωστή κατεύθυνση. Εδώ έχω κάποιες αμφιβολίες ό,τι αφορά την Τραπεζική Ένωση. Αυτά που ακούω ως αιτιολόγηση για την Τραπεζική Ένωση είναι ότι κάθε πολίτης στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να έχει την ίδια ασφάλεια για τις ε, αποταμιεύσεις του για τον τρίτο πυλώνα δηλαδή. Όμως αυτό μπορεί να επιτευχθεί και διαφορετικό, δηλαδή μπορεί να υπάρξει μια πανευρωπαϊκή διασφάλιση των καταθέσεων. Και αυτό μπορεί να γίνει και στη βάση κάποιου ανταγωνισμού. Να γίνει δηλαδή, δηλαδή, δηλαδή, δυνατό κάθε πολίτη στην Ευρώπη να έχει πρόσβαση σε κάθε τράπεζα. Ή κάθε τράπεζα να έχει τη δυνατότητα να δραστηριοποιείται σε κάθε χώρα μέλο. Τότε ο πολίτης είναι εκείνος ο οποίος θα αποφασίσει πλέον μόνο του που θα τοποθετήσει τα χρήματά του, ώστε να έχει τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Η ερώτησή μου προς εσά είναι, γιατί δεν προωθείτε μια τέτοια λύση στην βάση του ανταγωνισμού. Αντί υπέρ του έντις, που έχει ξεκάθαρα πολλά αδύνατα σημεία. Έχει μεγαλύτερο κίνδυνο, έχει μάλλον επιφέρει στρέβλωση του ανταγωνισμού ε, μεταξύ των τραπεζών μεταξύ αυτών δηλαδή που ανήκουν στην Τραπεζική Ένωση και αυτών που δεν θα ανήκουν στην Τραπεζική Ένωση και υπάρχει τελικός κίνδυνος. Ερώτηση λοιπόν, γιατί δεν προ... προτείνεται μια ανταγωνιστική λύση αφού ούτως ή άλλως η Ευρωπαϊκή Ένωση πολλά λέει υπέρ του ανταγωνισμού και της ανταγωνιστικότητας. Πολύ σύντομη δεύτερη ερώτηση. Είπατε ότι το Συμβούλιο ασχολείται με το πρόβλημα του ΦΠΑ χωρίς να δώσετε λεπτομέρειες. Θα ήθελα να μάθω, στο Συμβούλιο έχετε συζητήσει το ενδεχόμενο εισαγωγή reverse charge διαδικασίας, ενδεχομένως σε επίπεδο χωρών. Οι χώρες δηλαδή να αποφασίσουν αν θα κάνουν την reverse charge ή αν θα παραμείνουν στην διαδικασία standard charge. Um, thank you. Σας ευχαριστώ σχετικά με την ανταγωνιστικότητα στην Τραπεζική Ένωση είναι πολύ ενδιαφέρον. Αλλά εγώ νομίζω ότι κάθε φορά που ένας In whichever Σε κάθε, όπου και αν βρίσκεται εν πάση περιπτώσει ένας καταθέτης στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης αξίζει την ίδια προστασία. Βέβαια μπορεί να είναι ελεύθερο ο καθένα να επιλέξει το πιστοτικό ίδρυμα ή τη χώρα την οποία επιθυμεί και μπορεί επίσης να έχει την δυνατότητα να αλλάζει από πιστοτικό ίδρυμα σε πιστοτικό ίδρυμα. Και αυτό γίνεται και στη δική μου χώρα. Το σύστημα πάντως απαιτεί μεγαλύτερη διαφάνεια έτσι ώστε ο καταναλωτής να καταλάβει ποιες τράπεζες μπορούν να εμπιστευθούν, ποιες τράπεζες πρέπει να αντιμετωπίσουν με μεγαλύτερη επιφυλακτικότητα γιατί πολλές φορές οι καταθέτες δεν έχουν ε, καμία ιδέα γύρω από αυτά. Είναι δύσκολο να κατανοήσουν και να αξιολογήσουν τους κινδύνους και εδώ ακριβώς θα πρέπει να έχουμε ισχυρές εποπτικές αρχές, ε, ξεκάθαρες ε, νομοθετικές ρυθμίσεις, προστασία των επίπεδο κεφαλαίων προστασίας για τις τράπεζες, και έτσι το σύστημα θα είναι πολύ πιο ισχυρό και πιο ε, θα έλεγα χρήσιμο από ότι να υπάρχει ένα, ε, μια πολυδιάσπαση στα συστήματα αυτά. Πριν πάντως επιτρέψουμε ε, ας πούμε την κυρία Ντελάγκε να ενταχθεί στο δικό μας σύστημα ασφάλισης θα προσπαθήσουμε να δούμε τι κινδύνους η ίδια εμπεριέχει και αυτή είναι η συζήτηση ουσιαστικά την οποία κάνουμε. Υπάρχουν λοιπόν αρκετά επιχειρήματα έτσι ώστε να υπάρξει ένα κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασφάλειας, κοινό επαναλαμβάνω, αλλά παρόλα αυτά υπάρχουν κίνδυνοι στον πιστοτικό τομέα που δεν να, μπορούμε να αγνοήσουμε. Για τα ΦΠΑ υπάρχει μια συζήτηση η οποία γίνεται για το λεγόμενο reverse charge. Πολλές χώρες ε, υποστηρίζουν ότι πράγματι εμείς θα επιτρέψουμε σε κάποιες χώρες ή σε μία συγκεκριμένη χώρα για ένα πείραμα σε σχέση με το σύστημα αυτό. Δεν έχουμε αποφασίσει ακόμα, θα συζητήσουμε την επόμενη Παρασκευή. Θα πρέπει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας δώσει στοιχεία σε σχέση με τη λεγόμενη αντίστροφη χρέωση ή επιβάρυνση. Thank you. Ευχαριστώ πολύ, Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ που είστε εδώ. Είμαι εδώ, είμαι εδώ. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Ξέρουμε πόσο εκτιμούμε το γεγονός ότι έρχεστε εδώ για να έχουμε ανταλλαγή απόψεων. Ένα σχόλιο πρώτα απ' όλα. Το σχόλιο είναι ότι σας ευχαριστώ που πήρατε το λόγο για τις δηλώσεις του κυρίου Γιούγκερ επί της Γαλλίας ε, και σας το λέω ως Γαλλίδα γιατί μπορείτε να αξιοποιήσετε μόνο το άρθρο 6 της ε, διακήρυξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του 1989 που ε, ξεκίνησε στη Γαλλία, που λέει ότι ο νόμο πρέπει να είναι ίδιο για όλου. Αυτό είναι ένα από τα μεγάλα επιτεύγματα τη Γαλλική Επανάσταση. Γιατί να μην το αξιοποιήσετε. Πολύ συγκεκριμένη ερώτηση. Συμφωνείτε με τον κύριο Σόιμπλε που είπε ότι, ότι αν υπάρξει Brexit, το μέσα είναι μέσα και το έξω είναι έξω. Ο κύριος Ντέζελ. Αν συμφωνώ in is in και out is out. Ε, ναι, φυσικά. Γενικά συμφωνώ. Αλλά ας ξεκινήσω με θετικό τρόπο. Έχουν γίνει δύο δημοψηφίσματα στην Ολλανδία. Κάτι που δεν λειτουργεί είναι να απειλεί κανείς τους ψηφοφόρους και να τους πούν ε, τι άσχημο θα ήταν να επιλέξουν ε, κάποια επιλογή. Δεν νομίζω ότι είναι σωστή προσέγγιση. Τώρα βέβαια δεν ξέρω πώς ενδιαφέρονται για αυτά που λέω οι Βρετανοί ψηφοφόροι, αλλά εάν ενδιαφέρονταν θα έλεγα ότι υπάρχουν πολύ σωστά επιχειρήματα και ε, βάσιμα για την ευρωπαϊκή συνεργασία και είναι προς το βρετανικό συμφέρον για πολλούς λόγους. Νομίζω το βασικό θέμα στη συζήτηση για τον Brexit είναι η μετανάστευση. Αλλά δεν θα αποφύγετε τη μετανάστευση και τα προβλήματα εάν βγείτε από την Ένωση. Το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία θα εξακολουθήσουν να πρέπει να συνεργάζονται για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα στη μάχη. Θα πρέπει να συνεχίσουν να συνεργαζόμαστε και με την συμμετοχή των Βρετανών ε, για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα στην περιοχή της Τουρκίας, της Συρίας κτλ. Υπάρχουν πολύ σωστοί λόγοι γιατί χρειάζεται και για τους Βρετανούς η ευρωπαϊκή συνεργασία και για μένα. Δεν επαρκεί να παραμείνει απλώς ε, το Ηνωμένο Βασίλειο θα ήθελα να ξαναγίνουν ενεργό μέλος, να είναι στην πρωτοπορία του σχεδιασμού και εφαρμογή των αλλαγών. Όπως ήταν κάποτε. Αλλά τώρα έχουν γίνει όλο και περισσότερο παθητικοί, αμυντικοί. Αυτό που θα ήθελα είναι μια πολύ πιο ενεργή βρετανική παρουσία. Ο, η κυρία Γκουλαρόχη, όχι δεν είναι θέμα απειλής. Θέτω όμως ε, το θέμα εκατομμυρίων ενωσιακών πολιτών σε διάφορες ε, ε, χώρες μέλη που διαρωτώνται τι επιπτώσεις θα έχει το αποτελέσμα του δημοψηφίσματος για αυτούς. Αυτό εννοώ. Να μην εστιάζουμε μόνο σε μία χώρα, να μην αγνοούμε όλους τους άλλους. Παρουσιάσατε τους λόγους. Αλλά πρέπει να καταλάβετε ότι το γεγονό ότι ορισμένοι δεν μπορούν να επηρεάσουν την κατάσταση του δημιουργεί πολλού φόβου. Σωστό λέει ο κ. Ντάισεμπλουμ. Άψογα, λέει ο πρόεδρος. Δημήτρης Παπαδημούλης. I'll put my question in Greek, Mr. President. Ε, σας ευχαριστώ κύριε Ντάισεμπλουμ για την παρουσία σας εδώ. Αν δεν κάνω λάθος, τα τελευταία δύο χρόνια είναι η πρώτη φορά που ε, στην αρχική σας δήλωση δεν αναφέρεστε καθόλου στην Ελλάδα. Και αυτό το θεωρώ καλό σημάδι, όπως και το ότι η Ελλάδα έχει φύγει από τα πρωτοσέλιδα των διεθνών οικονομικών και πολιτικών ε, μέσων. Αλλά είσαστε και πρόεδρος του Eurogroup και σε δύο μέρες έχει συνεδρία στο Eurogroup. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω ε, τι αποφάσεις θα πάρετε στην Ελλάδα σε δύο μέρες, για την Ελλάδα σε δύο μέρες. Ε, θα δοθεί επιτέλους αυτή η δόση του δανείου και θα γίνει το αποφασιστικό βήμα για την ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης. Και η δεύτερη μου ερώτηση, πριν λίγες ημέρες, ε, ο κύριος Ντομπρόφσκης και ο κύριος Μοσκοβισή, μιλώντας στο Ευρωκοινοβούλιο, είπαν ότι είναι αισιόδοξοι ότι αμέσως μετά το καλοκαίρι θα προχωρήσουν οι συζητήσεις ανάμεσα στους δανειστές, τους Ευρωπαίους δανειστές και το IMF προκειμένου να συγκεκριμενοποιηθεί ο οδικός χάρτης για την ελάφρυση του χρέους. Σημερίζεστε αυτή την εκτίμηση. Και επίσης ο κύριος Ντομπρόφσκης είπε ότι για μετά το 2018 εξετάζει η Κομισιόν χαμηλότερα, ρεαλιστικότερα πρωτογενή πλεονάσματα σε σχέση με το 3,5% που σχεδόν οι πάντες το θεωρούν ανέφικτο να διατηρηθεί για μια δεκαετία. Χτες μόλις στους Financial Times ο κύριος Τουρνάρας, διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας και πρώην υπουργό Οικονομικών, υποστηρίζει ότι θα πρέπει και οι δανειστές να συντρέξουν έτσι ώστε χωρίς καθυστερήσεις να υπάρξει επιτέλους αυτή η ελάφρυση του χρέους την οποία ζητάει και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προκειμένου να συμμετάσχει και χαμηλά πρωτογενή πλεονάσματα από το 18 και μετά της τάξης του 1,5 έως 2% αντί για 3,5 προκειμένου να επιστρέψει η Ελλάδα με ένα βιώσιμο και σταθερό τρόπο στην ανάπτυξη και να δοθεί ένα σήμα στους επενδυτές και στις αγορές ότι μπαίνει σε μια περίοδο κανονικότητας η, η, χώρα μου. Πώς απαντάτε σε αυτές τις ιδέες. Thank uh, Σας ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας. Εγώ είμαι εδώ σαν πρόεδρος του ΕΚΟΦΗΝ, οπότε δεν θα απαντήσω για το Eurogroup. Θα μπορούσα να το πω. Απλά θα σας δώσω απλές απαντήσεις. Έχετε δίκιο. Εγώ δεν αναφέρθηκα στην Ελλάδα. Ο επίσημος λόγος είναι ότι είμαι εδώ για το ΕΚΟΦΗΝ. Υπάρχει κι άλλος ένας λόγος, τον οποίο είπατε εσείς. Βρισκόμαστε σε μια διαφορετική φάση τώρα. το μέγεθος της εμπιστοσύνης ανάμεσα στην Ευρωζώνη, στα υπόλοιπα μέλη και στην Ελλάδα είχε πέσει πάρα πολύ το προηγούμενο καλοκαίρι. Το βιώσαμε αυτό και από τότε τα πράγματα έχουν αλλάξει, έχουν αλλάξει πολύ, υπάρχει μια διαφορετική ατμόσφαιρα, δουλεύουμε επικοδομητικά, υπάρχουν διαφορές φυσικά, υπάρχουν διαφορές για το ποιος είναι ο σωστός δρόμος, αλλά πάντως επικοδομητικά συνεχίζουμε να δουλεύουμε και γι' αυτό ακριβώς νομίζω ότι και στα πλαίσια ακριβώς των υπευθύνων του ESM να δώσουμε την άδεια και ε, για την... Ε, Prior uh, ε, Για την επόμενη δόση. Λοιπόν, τώρα για τα θέματα αν θα υπάρξει συζήτηση για το χρέος μετά το καλοκαίρι άμεσα. Κοιτάξτε, δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο. Υπάρχει ο λεγόμενος οδικός χάρτης εμείς έχουμε πει πώς θα αντιδράσουμε στο θέμα του χρέους, στη συμφωνία την οποία, στην οποία καταλήξαμε τον προηγούμενο μήνα. Το ESM θα δει ακριβώς πώς θα προχωρήσουμε στο θέμα της διαχείρισης του χρέους, να μειώσουμε τα επιτόκια, να διαχειριστούμε με πιο ευνοϊκό τρόπο το χρέος τα επόμενα χρόνια. Αυτά τα μέτρα μπορούν να ληφθούν εκ των προτέρων. Στο τέλος του προγράμματος Έχουμε άλλες δυνατότητες, άλλα μέτρα από τα οποία μπορούμε να πάρουμε. Θα δούμε ακριβώς τι θέματα τίθενται σε σχέση με τη βιωσιμότητα εκείνη τη στιγμή. Και για την επόμενη περίοδο, αν χρειαστεί θα κάνουμε και περισσότερα. Το κομβικό ερώτημα το οποίο αυτή τη στιγμή τέθηκε από τον κύριο Στουρνάρα είναι το πλεόνασμα 3,5% για το 18, αν κάτι τέτοιο είναι ρεαλιστικό ή μήπω είναι ιδιαίτερα υψηλό. Εμείς συμφωνήσαμε ότι αυτό το 3,5% για μια μακρά περίοδο δεν είναι κάτι το ρεαλιστικό. Έχουμε βάλει λοιπόν από το 3,5% να κατεβαίνει την επόμενη, τις επόμενες δεκαετίες. Αλλά παρόλα αυτά δεν τίθεται το θέμα τώρα. Στο τέλος του χρόνου, όταν το ΔΝΤ θα παρουσιάσει την δική του απόφαση, την απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου. Ε, θα περιμένουμε την απόφαση αυτή και θα δούμε από εκεί και πέρα τι θα κάνουμε. Thank you, Philip Ο κύριος Λάμπερτ. Κύριε, κύριε Ντάσελμπου, καλή σας μέρα. Η Ολλανδική Προεδρία είχε μεγαλύτερες ελπίδες από αυτές που τελικώς ε, φάνηκε να υλοποιούνται. Βεβαίως, η Προεδρία δεν έχει τα πάντα στα χέρια της. Για το έντις μου φαίνεται το έκοφιν να θέλει να στείλει την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξανά στην φάση του σχεδιασμού. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι ευαίσθητο το θέμα αυτό και πρέπει να προχωρήσουμε προσεκτικά δεν ε, τρέχει η δουλειά ούτε εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο με μεγάλη ταχύτητα. Όμως όταν μιλείτε για το 2024 κάπως ανησυχώ. Σχετικά δηλαδή με, το, με τη δέσμη μέτρων για την φόρο αποφυγή, ο, όσα ήδη δεν κάλυψε όλα τα θέματα. Αποδυνάμωσε λοιπόν τα ε, μέτρα του ΩΣΑ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τώρα το ΕΚΟΦΗΝ αποδυναμώνει και αυτά της Επιτροπής αναρωτιέμαι τι θα μείνει στο τέλος από τη φιλόδοξη αυτή ατζέντα. Και έχω την εντύπωση ότι υπάρχουν άλλοι που έχουν μεγαλύτερη βαρύτητα από εσάς, από τον κύριο Ντάισερμπλουμ δηλαδή. Ποιος είναι αυτός? Έρικ Λίβες, ο συνάδελφός σας, υφυπουργός οικονομικών. Γνωρίζετε για ποιον μιλώ. φαίνεται πως κυριαρχεί περισσότερο η άποψή του από τη δική σας. Τώρα, για τους κανόνες. Εάν έχουμε κανόνες και θέλουμε να γίνονται σεβαστοί, πρέπει να εφαρμόζονται. Όμως, από την άλλη μεριά, εάν οι κανόνες έχουν σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο που τελικώς θα παράγουν το αντίθετο αποτέλεσμα, τότε πρέπει να αναρωτηθούμε αν οι κανόνες είναι σωστοί. Όχι αν χρειάζονται κανόνες, αλλά αν οι κανόνες αυτοί είναι οι σωστοί. Και είμαι πεπισμένος ότι οι κανόνες οικονομικής διακυβέρνησης επιτείνουν την κυκλική κίνηση και αντί να το λαμβάνουμε αυτό υπόψη, στην πραγματικότητα προσφέρουμε σε αυτούς πολύ μεγάλη διακριτική ευχαίρεια για το τι θα κάνουμε. Ξαναλέω, αν δεν εξυπηρετούν το στόχο τους οι κανόνες, ας τους αλλάξουμε. Όχι να λέμε ότι α, πιστεύουμε στους κανόνες αυτού, αλλά δεν του εφαρμόζουμε. Τι, ποια είναι η απόψή σα. Ευχαριστώ κύριε Λάμπερτ. Αυτά που μου είπατε μου φαίνεται, εγώ τα δέχομαι ως φιλοφρόνηση. Διότι είπατε ότι αναμένατε πολύ περισσότερα από την Ολλανδική Προεδρία. Εμεί προσπαθούμε να υλοποιήσουμε, δηλαδή να σας ικανοποιήσουμε. Μα μένουν λίγε μέρε ακόμη, ίσως προλάβουμε να βελτιώσουμε τον τελικό βαθμό που θα μας βάλετε. Για το ΕΔΙΣ λέτε ότι στέλνουμε την Επιτροπή ξανά στη φάση του σχεδιασμού, να τα ξανασχεδιάσει. Δεν νομίζω την αλήθεια αυτό. Μιλούμε για το roadmap αυτό και ποια βήματα θα κάνουμε τα επόμενα χρόνια. Όμως η τεχνική εργασία γίνεται και στο επίπεδο του Συμβουλίου πάνω στην πρόταση έντις. Το Συμβούλιο δηλαδή έχει αναλάβει τώρα την επεξεργασία της προτάσεως Θα αλλάξουν πράγματα στη διαπραγματεύση. Ναι, βέβαια, πάντα γίνεται αυτό. Όχι όμως στέλνοντας την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξανά στο τραπέζι του σχεδιαστή. σας ανησυχεί, λέτε, το 2024. Εμένα όχι. Έχει συμφωνηθεί και μεταξύ μας και των κοινοβουλίων δηλαδή. Και το, ε, το Ταμείο για την εξηγήση των Τραπεζών θα πρέπει και αυτό να είναι έτοιμο μέχρι το 2024. Έχει καλώς λοιπόν μέχρι τότε, άρα η Τραπεζική Ένωση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί. Αυτό όμως απαιτεί και άλλα στοιχεία. Αυτά τα οποία έχουμε ήδη καταγράψει, με ποιο τρόπο θα τα χειριστούμε, πώς θα πετύχουμε τις πολιτικές ισορροπίες και όλο αυτό θα συναποτελέσει τον οδικό χάρτη. Τέλος, λέτε ότι είστε απογοητευμένο σχετικά με την φορά φοροαποφυγή. Δώστε μας τουλάχιστον μια ευκαιρία. Θα μπορούσα να είχα πετύχει συμφωνία για την ATAD, για τη σχετική οδηγία δηλαδή, ήδη από τον προηγούμενο μήνα στο Συμβούλιο. Όμως, θα έπρεπε να είχα κάνει μεγάλες παραχωρήσεις, διότι οι υπουργοί μου λένε «Α, θέλουμε αυτό, δεν θέλουμε εκείνο». Μπορώ να τα δεχτώ όλα αυτά, τους είπα, και μετά να βγω από την αίθουσα και να πω «Α, πετύχαμε συμφωνία», αλλά τελικά τα χέρια μου θα είναι άδεια. Αφήστε λοιπόν να συνεχίσουμε να ε, διαπραγματευόμαστε. Ούτως ή άλλω η αλλω η Ένωση βρίσκεται ε, ε, σε πρωτοπόρα θέση σε ό,τι αφορά τα BEPS παγκοσμίω. Τώρα, αν νομίζετε ότι οι κανόνε παράγουν το αντίθετο αποτέλεσμα, τότε πράγματι να του αλλάξετε. Είναι σωστή η συζήτηση αυτή στο άτυπο συμβούλιο ΕΚΟΦΗΝ στο Άμστερνταμ συζητήσαμε σχετικά με το πώς λειτουργούν τώρα οι δημοσιονομικοί κανόνες. Για παράδειγμα, ο, ο δείκτης διαστοτικού ελλείμματος. Πώς λειτουργεί και πώς επιτρέπει να προβλέψουμε και πώς μπορούν, πώς μπορούν πολιτικά να το επηρεάσουν. Θα έρθει λοιπόν να υποβάλει προτάσεις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αργότερα φέτος για να αλλάξουν οι δείκτες για το σύμφωνο και ιδίω για το προληπτικό σκέλος. Όντω, ίσω πρέπει να αλλάξουμε του κανόνε, ίσω όντω να μην αποδίδουν. Όμω, αν έχετε κανόνε, καταθέτετε νομοθετικέ προτάσει και εκεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πληρεί απολύτω τον ρόλο τη. Χρησιμοποιεί δευκαμψία και οτιδήποτε άλλο έχει στην εργαλειοθήκη τη. Έχει καλώ. Όμω, με τρόπο αντικειμενικό. Συμφωνώ μαζί σας όμως σε αυτό που λέτε εν κατακλείδη εάν έχετε κανόνες και δεν σας αρέσουν αλλάξτε τους και τότε εφαρμόστε τους αλλαγμένους. Να το πω αυτά που λέτε, μπορώ να τα χρησιμοποιήσω, λέει ο πρόεδρος, ωραία. Μάρκο Βάλλη. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ τον Ολλανδό Υπουργό λοιπόν που είναι μαζί μας σήμερα. Μιλήσατε για ένα οδικό χάρτη. Είναι πολύ της μόδας αυτό. Για ένα οδικό χάρτη τον οποίο συνέγραψαν πέντε πρόεδροι, όπως λέγεται η ομάδα αυτή, Μιλάμε για την Τραπεζική Ένωση, ο κόσμος θέλει μια Τραπεζική Ένωση η οποία δεν θα επιτρέπει καταχρήσει στον τομέα ακριβώς τον χρηματοπιστωτικό όπως έχει η κατάσταση και οι προτάσεις αυτές φοβάμαι ότι θα μεγενθύνουν το πρόβλημα και τα νέα πιστοτικά προϊόντα δεν είναι επαρκώς διαφανή έτσι ώστε και εσείς προσπαθήσατε να τα μετατρέψετε, να κάνετε την κατάσταση κάπως καλύτερη αλλά δεν διορθώνονται τα πράγματα στο θέμα της προστασίας των καταθέσεων. Υπάρχει μία μείωση του κινδύνου αλλά νομίζω ότι γίνεται με λάθος όρους. Ε, υπάρχει η έκθεση στο δημόσιο χρέος, είναι κάτι το οποίο ε, θα έλεγα δεν είναι του ιδίου επίπεδου ε, με τα προβλήματα που δημιουργούνται σε επίπεδο συναλλαγών ανάμεσα σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα αγνοείται η βούληση του λαού και γίνεται δεκτή και ακούγεται η δύναμη των λόμπι και των τραπεζών. Και υπάρχει και η μεγάλη φοροδιαφυγή επίσης. Ξέρετε ότι υπάρχουν ακόμα χώρες που έχουν θέσεις διαφορετικές με την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Κοινοβουλίου για το πακέτο που προετοιμάζουμε. Ε, η Ολλανδία είναι υπέρα αλλά υπάρχουν άλλες χώρες οι οποίες είναι κατά και πάντα για τον οδικό χάρτη των πέντε προέδρων μετά από το Brexit και τα λοιπά υπάρχει ένας οδικός χάρτης σχετικά με τις δημοσιονομικές δυνάμεις της Ευρωζώνης. Τι θα γίνει μετά. Ο κόσμος προσπαθεί να μάθει. Στην Ευρώπη εμείς έχουμε μπροστά μας το πρόβλημα το οποίο δημιουργεί επίσης η Γερμανία και το πλεόνασμά της το οποίο καταστρέφει την εσωτερική αγορά. Θα ήθελα να μάθω αν οι δημοσιονομικές αυτές δυνατότητες της Ένωσης θα μπορέσουν να αντιμετωπιστούν με καλύτερο τρόπο από πλευράς της ε, Γερμανίας. Ε, δύσκολα μου βάζετε κύριε Βάλλη. Ε, Κυρίω γιατί δεν καταλαβαίνω, δεν είμαι σίγουρο ότι καταλαβαίνω. Είπατε ότι η Τραπεζική Ένωση θα οδηγήσει σε νέα χρηματοπιστωτικά προϊόντα με ωραία ονόματα. Τι ακριβώ εννοείτε, δεν καταλαβαίνω. Είπατε ότι βασιζόμαστε σε λάθος ε, κριτήρια. Για την ε, Ένωση Κεφαλαίου λέει ο κύριος Βάλλη. Mm, λέει ο κύριος Νομίζω ότι η ερώτησή σας τελικά ήταν αν θα ακούσετε μόνο τις τράπεζες ή τους πολίτες. Νομίζω ότι οι πολίτες ενδιαφέρονται οι τράπεζές τους να είναι ασφαλείς, να έχουν εμπιστοσύνη στις τράπεζές τους και τις οποίες δεν χρειάζεται να διασώζουν ε, κάθε λίγο και λιγάκι με τα χρήματά τους ε, των φορολογουμένων ε, με τεράστιο κόστος τρομερή αύξηση του δημοσίου χρέου. Και ήταν ένα από του λόγου για του οποίου χρειάστηκε να διασωθούν οι τράπεζε. Βεβαίω πρέπει να δούμε τι κίνδυνοι υπάρχουν στο τραπεζικό μα σύστημα και να αντιμετωπίσουμε αυτού του κινδύνου με λογικό και σταδιακό τρόπο. Ούτω ώστε οι τραπεζέ μα να είναι υγιεί, ισχυρέ, ε, να μπορούν να αντιμετωπίσουν του κινδύνου που δημιουργούν μόνες τους και να είναι ε, σε θέση να διανοηδιωτήσουν τις επιχειρήσεις και τους ε, καταναλωτές. Τελεία. Για το ή για το φόρο. Με ρωτήσατε ποιες χώρες ε, αντιτίθενται. Ποτέ δεν λέω ποιες χώρες είναι υπέρ κατά. Αυτό που μετράει σε τελευταία ανάλυση από πλευράς Προεδρίας είναι να καταλήξουμε σε συμφωνία και σε μια συμφωνία που να είναι όσο δυνατόν ισχυρότερη και αποτελεσματικότερη. Και είμαστε ε, στα πλαίσια αυτής της διαδικασίας να προσπαθήσουμε να συμφωνήσουν για τα διάφορα θέματα όλες οι χώρες. Τέλος, Αναφερθήκατε στο ότι η Γερμανία έχει μεγάλο πλεόνασμα. Μα δεν είναι η μόνη χώρα που έχει μεγάλο πλεόνασμα. Ευχαριστώ πολύ. Αλλά δεν κατάλαβα τι σχέση έχει αυτό με την ε, φορολογική ικανότητα της Ένωσης. Όταν δεν καταλαβαίνω τις ερωτήσεις ε, δυσκολεύομαι να απαντήσω. Όχι, όχι, παρακαλώ, δεν έχουμε χρόνο, λέει ο κύριος ε, Κύριε Υπουργέ Οικονομικών της Ολλανδίας, στα πλαίσια της ε, Ευρωπαϊκής Οικονομικής Διακυβέρνησης θα σας μιλήσω για τα δημοσιονομικά της χώρας μου και της χώρας σας. Ε, με εκνεύρισαν λιγάκι οι δηλώσεις που κάνατε στα, σε διάφορα άρθρα και σε μια συνέντευξη στο Φιγκαρό αρχές Ιουνίου Είπατε ότι είναι απαράδεκτη η επιοίκεια της, ε, των Βρυξελών έναντι της Γαλλίας και ότι είναι απαράδεκτο και χάνει αξιοπιστία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν δεν επιβάλλει τους ε, κανόνες, για παράδειγμα το 3% του ελλείμματος. Ενώ η γαλλική κυβέρνηση προσπαθεί να πάρει 1,6 δις από την Google που ε, απειλείται και για χρόνια δεν έχει πληρώσει φόρο ακριβώς επειδή εποφελείται από τους ευνοϊκούς κανόνες ε, της ε, Ολλανδίας και η Γαλλία δεν είναι το μόνο θύμα αυτής της φορολογικής πολιτικής της κυβέρνησής σας και δεν είναι η μόνη επιχείρηση Google που έχει ωφεληθεί. Για τη Γαλλία το έλλειμμα κέρδους ε, είναι 30 με 40 δις το χρόνο που είναι 2% του ΑΕΠ. Οι επενδύσεις που περνάνε από την χώρα σας είναι οικονομικές ροές που φεύγουν από άλλες χώρες. Έχουμε μια έκθεση από το δικό μας κοινοβούλιο που λέει ότι έχουμε μεγάλες δυσχέρειες στη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων και πρέπει να επιβάλλουμε αυτήν την ε, λιτότητα που είναι τόσο σκληρή για τους λαούς. Και Εν τω μεταξύ, οι πολυεθνικέ επενδύουν σε φορολογικού παραδείσους ε, τα απαράδεκτα κέρδη που έχουν από τη χώρα πώς Πώ τολμάτε να δίνετε μαθήματα στη χώρα μας ενώ οι διαδοχικέ σας κυβερνήσεις εδώ και δεκαετίες έχουν συμβάλει στην ε, μείωση των εσόδων τη χώρα μου. Είναι απαράδεκτη αυτή η τακτική σας. Το έλλειμμά μας 3,5 του ΑΕΠ θα ήταν μόνο 1,5 το πολύ εάν δεν υπήρχαν ορισμένε χώρε που έχουν κάνει ε, επιχείρηση την ε, φόρο απαλλαγή. Οι φόροι που δεν πληρώνουν οι πολυεθνικές στη Γαλλία προκαλούν τα ελλείμματα για τα οποία μας κατηγορείτε και ε, επίσης προκαλούν τη λιτότητα που μας επιβάλλεται. Γιατί λοιπόν θα πρέπει να ακούσουμε τις επικρίσεις ενός υπουργού μιας χώρας που είναι συνένοχος σε σοβαρά φορολογικά εγκλήματα. Σας ευχαριστώ πολύ για την απάντησή σας. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο κ. Ντάζεμπλουμ. Και πρώτα, οι παρατηρήσεις μου σχετικά με το ρόλο της Επιτροπής για το ε, σύμφωνο είχε ελάχιστα, ε, ελάχιστα να κάνουν με την Γαλλία. Εγώ δεν σχολίασα την περίπτωση της Γαλλίας, αλλά την περίπτωση συγκεκριμένων αποφάσεων. Δόθηκαν κάποια χρόνια στη Γαλλία για να μειώσει το έλλειμμά τη και αυτό μπορεί να είναι πολύ θετικό αντικειμενικά. Και σε άλλε χώρε δόθηκαν παραπάνω χρόνια για να αντιμετωπίσουν τα έλλειμματά του και να συμμορφωθούν ξανά με το σύμφωνο. Δεν έχω πρόβλημα εφόσον αυτό γίνεται στην βάση διαφανών και αντικειμενικών κριτηρίων. Αυτό έλεγα στις παρατηρήσεις μου. Για την φοροδιαφυγή, μάλιστα αυτό συμβαίνει και το γνωρίζουμε όλοι μας. Έχω ξαναπεί ότι εάν οι κάτω χώρες υπήρξαν τμήμα του προβλήματος έως τώρα και υποθέτω ότι είμαστε, τότε θα πρέπει να αποτελέσουμε μέρος της λύσεως. Και αυτή είναι και η θέση που έχω και ως πρόεδρος του Eurogroup αλλά και ως Υπουργός Οικονομικών. Το φορολογικό μας σύστημα επέτρεψε σε διεθνείς εταιρείε να αποφύγουν την καταβολή φόρων, όχι μόνο μέσω Ολλανδίας. Αν είχαμε πολλοί αυτούς κανόνες θα είχαν πάρει άλλη διαδρομή. Υπάρχουν πολλέ χώρες που έχουν τέτοιους κανόνες. Χρειάζονται διεθνή στάνταρτ, χρειάζεται να εφαρμόζονται σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό ακριβώς πάμε να κάνουμε. Εάν αυτό απαιτήσει τροποποίηση τη νομοθεσία στη δική σας χώρα ή στη δική μου χώρα, α το κάνουμε. Εμείς πάντως θα το κάνουμε. Ήδη φέτος θα αλλάξουμε την νομοθεσία μα, για παράδειγμα, για το λεγόμενο Innovation Box. Ένα από τα εργαλεία που είχαν φορολογικά εργαλεία δηλαδή, που είχαν κάνει τι κάτω χώρε πάρα πολύ ελκυστικέ για ε, αλλοδαπές εταιρείε. Νομίζω όμω ότι αυτό είναι ο μόνο δρόμο προ τα εμπρό. Χρειάζονται λοιπόν πολύ ξεκάθαρα διεθνή στάνταρτ που θα εφαρμόζονται σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνική νομοθεσία για να σταματήσουν αυτά που επισημάνατε. Και εγώ είμαι αποφασισμένο να το πράξω. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρο Γκουαλτιέρη. Ο κ. Αριανόπουλο. Η ερώτησή μου, σαν αφορμή έχει μονάχα την κατάσταση στην Ελλάδα, αφορά ολόκληρη την Ευρώπη, όπως δείχνουν και οι κινητοποιήσεις των εργαζόμενων στη Γαλλία και σε άλλες χώρες. Και μάλιστα με αφορμή αυτό το οποίο υπόθηκε από την εισήγηση, ότι επεξεργάζεται η Επιτροπή ενιαίους κανόνες για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση για τον καθορισμό των μισθών με βάση την ανταγωνιστικότητα. Κύριε Ντάισελμπλουμ, δώσατε συγχαρητήρια και εσείς προσωπικά και ο κύριος Σόιμπλε και ο Πρωθυπουργό τη Γαλλία, τον κύριο Τσίπρα και στην κυβέρνησή του για τι μεταρρυθμίσει που έκανε για να, κατά τη διάρκεια τη πρώτη αξιολόγηση. Βέβαια, συγχαρητήρια δεν του δίνει ο λαό, διότι για 14η φορά μειώνονται οι συντάξει, οι μισθοί, έχουν εκτοξευθεί οι φόροι όσον αφορά το λαό, ετοιμάζονται χιλιάδε κατασχέσει σπιτιών από τι τράπεζε, οι οποίε μάλιστα δίνουν τα κόκκινα δάνεια στα, ε, στα κτλ. Και ενώ είστε τόσο περιοριστικοί όσον αφορά το εισόδημα το λαϊκό, είστε ιδιαίτερα γαλαντόμοι και εσείς και η κυβέρνηση όσον αφορά το τι θα δώσετε προνόμια, επιδοτήσει και φοροαπαλλαγές στι μεγάλε επιχειρήσει, με τον νέο αναπτυξιακό νόμο τον οποίο έχετε εγκρίνει και εσεί. Επειδή λοιπόν μπαίνετε σε καινούργια διαπραγμάτευση για τη δεύτερη αξιολόγηση για το επόμενο φθινόπωρο και ο λαός ανησυχεί γιατί κάθε διαπραγμάτευση τον φτωχαίνει ακόμα περισσότερο, έχω να σας κάνω ορισμένες πολύ συγκεκριμένες ερωτήσεις και θα ζητούσα πολύ συγκεκριμένε απαντήσει. Επειδή είναι γνωστό ότι θα συζητήσετε με την ελληνική κυβέρνηση το λεγόμενο εργασιακό πακέτο. Τι εννοείτε όταν λέτε βέλτιστε πρακτικέ, το οποίο περιλαμβάνεται και στο τρίτο μνημόνιο με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Εννοείτε την απελευθέρωση των ομαδικών απολύσεων, γιατί αυτό συζητάτε, ιδιαίτερα μάλιστα μετά από την εισήγηση του εισαγγελέα του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που λέει ότι πρέπει να απελευθερωθούν οι ομαδικές απολύσεις και να γίνει κόλαση σε μια χώρα που έχει ήδη 25% ανεργία και δεν μειώνεται παρά τα μέτρα που παίρνετε. Δεύτερον, τι εννοείται βέλτιστε πρακτικέ για του μισθού και νέο σύστημα μισθών. Γιατί σήμερα γράφεται στον τύπο αυτά τα οποία συζητούνται, δηλαδή να κατεργηθει 13 13ο και 14ο μισθό να μειωθεί ακόμα περισσότερο ο κατώτερος μισθός κάτω από 586. Και τελείωσα, τελείωσα. Και να υπάρχει, να υπάρχει μόνιμος, μόνιμος αμετάβλητος μισθός στην εργασία σου και τέλος. Um, Πολύ συγκεκριμένες ερωτήσεις και χρειάζονται πολύ συγκεκριμένες απαντήσεις τι οποίες δεν μπορώ να δώσω τώρα για τι μεταρρυθμίσει στην αγορά εργασία. Ε, μόλις έχουν ξεκινήσει. Στο τέλος της διαδικασίας αυτής, έτσι όπως προβλέπονται, οι θεσμοί θα ενημερώσουν και τους υπόλοιπους ε, ε, υπουργούς στο Eurogroup, συνεπώς δεν μπορώ να σας δώσω λεπτομέρειες σε σχέση με τις ερωτήσεις που θέσατε. Γκούνα Χακμακ, ευχαριστώ πολύ. Θέλω να θέσω ένα θέμα για το συνολικό γενικό οικονομικό κλίμα. Γιατί μου δημιουργήθηκε κάπως η εντύπωση ε, που αυτό που εννοώ τώρα είναι και μία δική μου απογοήτευση είναι ότι συζητάμε διαρθωτικές μεταρρυθμίσεις. Όταν υπάρχει ένα διαρθωτικό πρόβλημα, συζητάμε, δημιουργούμε μια νέα επιτροπή, καθορίζουμε ένα νέο οδικό χάρτη ε, και ε, ορισμένους ε, νέους κανόνες που δεν τους εφαρμόζουμε, τους αντικαθιστούμε με νέους νόμους που ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να τους εφαρμόζουμε. Να τους εφαρμόσουμε, αλλά δεν αλλάζει η κατάσταση. Και αν δούμε την ευρωπαϊκή οικονομία συνολικά από το 2007 και μετά, οι άμεσες ε, ε, εξωτερικές επενδύσεις έχουν πέσει στο 50% περίπου. Αυτή είναι η συνολική εικόνα. Ενώ για άλλες περιοχές του κόσμου έχουν αυξηθεί, έχουν διπλασιαστεί προς τις ΗΠΑ. Έχουμε λοιπόν έλλειμμα επενδύσεων. Το πρόβλημα που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το φορολογικό βάρος είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση 10 με 15% υψηλότερο από οποιαδήποτε άλλη περιοχή του κόσμου που μας ανταγωνίζεται. Διερωτώ με τι πρέπει να κάνουμε, δηλαδή για να έχουμε ένα θεματολόγιο διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, να κάνουμε περισσότερη προσπάθεια για να αλλάξουμε ακριβώς τις προϋποθέσεις για τη λειτουργία της οικονομίας και όχι να συζητάμε αυτό που μας ενδιαφέρει περισσότερο, πώς να αλλάξουμε τα θεσμικά όργανα της Ένωσης. Γιατί καμία από αυτές τις αλλαγές δεν θα προκαλέσει αυτομάτως διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Τι θα κάνουμε λοιπόν για να συζητήσουμε συνολικά την ευρωπαϊκή οικονομία και όχι τα ευρωπαϊκά όργανα και επιτροπές. Ο κύριος Ντάιζελ, ευχαριστώ, έχετε απόλυτο δίκιο. Ε, αφιερώνουμε υπερβολικά πολύ χρόνο σε θεσμικά θέματα. Πιστεύω ότι εξακολουθούν οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις να είναι το κύριο θέμα για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και για να επιτύχουμε υψηλότερη ανάπτυξη. Δεν μπορούμε να αποδεχθούμε το σημερινό πολύ χαμηλό επίπεδο ανάπτυξης σε σχέση ακριβώς και με τα ποσοστά ανεργίας. Πρέπει λοιπόν να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες που υπάρχουν ακόμη περισσότερο για εμβάθυνση της εσωτερικής αγοράς. Να δημιουργήσουμε περισσότερες δυνατότητες επενδύσεων σε διάφορους κλάδους της οικονομίας μας. Και γι' αυτό ο Πρωθυπουργός μου μαζί με τον Πρόεδρο Γιούνκερ έγραψαν ένα άρθρο, πιστεύω, στην εφημερίδα Financial Times, τονίζοντας ιδιαίτερα την ανάγκη ολοκλήρωσης της ε, εσωτερικής αγοράς. Υπάρχει πολύ δυναμικό ανάπτυξης ε, αν το κάνουμε αυτό και δεν καταλαβαίνω γιατί το υποτιμούμε. Το πρόγραμμα Juncker είχε τρεις πυλώνες αν θυμάστε και ο τρίτος έλεγε ότι πρέπει να δημιουργήσουμε περισσότερες δυνατότητες επενδύσεων μέσω διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και δεν έχει επιτευχθεί επαρκής πρόοδο. Ε για το θέμα αυτό. Και το ίδιο ισχύει και για αυτό που είπατε ότι είναι πολύ υψηλή η φορολογική επιβάρυνση. Αν δείτε πολύ λειτουργούν οι αγορές εργασίας, έχουμε ένα πολύ ρωμαλαίο κοινωνικό πρότυπο στην Ευρώπη που ως σοσιαλδημοκράτης ε, το εκτιμώ ιδιαίτερα, αλλά το κόστος τελικά βαραίνει ιδιαίτερα το λιγότερο παραγωγικό κομμάτι της οικονομίας μας. Πρέπει λοιπόν να γίνει ανακατανομή του φορολογικού βάρους για να μπορούμε να δημιουργούμε δυνατότητες ε, πρόσληψης των εργαζομένων. Είναι σημαντικές μεταρρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν σε όλες τις χώρες. Οι υπηρεσίες σε πολλές ε, χώρες ε, είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό ακόμη υπερβολικά έχουν πολύ υπερβολικούς κανόνες υπάρχουν πολλά κλειστά επαγγέλματα υπάρχει πολύ γραφειοκρατία είναι πολύ δύσκολο για τους νέους να ξεκινήσουν επιχειρήσεις Συμφωνώ. Πρέπει να τα κάνουμε όλα αυτά και πολλέ δυνατοτικέ μεταρρυθμίσει φυσικά δεν είναι δημοφιλεί και όλοι ω πολιτικοί προσπαθούμε να κερδίσουμε τι επόμενε εκλογέ. Αλλά αν δεν τι κάνουμε αυτέ τι μεταρρυθμίσει, τότε η οικόνομη θα μείνει σε αυτόν τον πολύ χαμηλό ρυθμό ανάπτυξη. Οπότε και η πιθανότητα να κερδίσουμε τι επόμενε εκλογέ θα παραμείνει εξίσου μικρή. Ευχαριστώ, Πολ Τάνγκ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ελπίζω ότι θα ολοκληρώσουμε την ΑΕΟΠΑ τούτη την εβδομάδα. Είμαι κάπως επιφυλακτικό σχετικά με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πάντως έχουμε επιτελέσει σημαντική πρόοδο και ελπίζω να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε μέχρι την Τετάρτη. Και να πούμε ότι έχουμε βελτιώσει την πρόταση που είχε κατατεθεί. και ότι έχουμε βάλει και κάποια τάξη στο χάος των διαμεθοριακών ε, συναλλαγών. Ερώτηση. για την φόρο αποφυγή. Το Κοινοβούλιο ενέκρινε την έκθεση Μπαγέτς που λέει ότι, και αυτό δείχνει μάλλον ότι με παρόλες τις μεγάλες πολιτικές διαφορές μπορούμε να συμφωνήσουμε πάνω σε μια συστημική προσέγγιση κατά της φοροαποφυγής. Υπάρχουν βέβαια διαφορές, μπορείτε να πείτε κάτι σχετικά, διότι φοβούμε ότι οι χώρες μέλη λένε τώρα ναι αλλά μετά κάνουν άλλα πράγματα. Όταν διαβάζω για παράδειγμα ότι η Ιρλανδία είναι αντίθετη με τις πληκτρινόμενες αλλαγές στο COC, βλέπω τον Σόιπλε να απειλεί ότι θα αφήσει το μισό πακέτο. Αυτά είναι άσχημα νέα. Μπορείτε να μας πείτε περισσότερα σχετικά με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζετε για το θέμα αυτό. Ο κύριος θα γίνει πολύ δυσκολότερη η ζωή μου αν σε πολλές λεπτομέρειες και σχετικά με τις διάφορες ενστάσει απέναντι στις διάφορες προτάσεις. Προτιμώ να παραμείνει το πακέτο ισχυρό και αξιόπιστο μέχρι τέλους της προσπάθειας. Δεν θέλω να βγω από την αίθουσα με κάτι που θα είναι αποδυναμωμένο και θα στερείται αξιοπιστία. Όλες, σε, όλες, σε όλες τις χώρες μας γίνονται τεράστιες συζητήσεις αυτή τη στιγμή σχετικά με τη αποφυγή, με την αδικία που προκαλεί η αποφυγή και ούτω καθεξής. Και όλοι μας οι Υπουργοί Οικονομικών στο ΕΚΟΦΗΝ οφείλουμε να συνεργαστούμε για να σταματήσει αυτό. Αν θέλουμε οι πολίτες και οι εταιρείε να πληρώνουν φόρους, αυτοί οι φόροι θα πρέπει να είναι δίκαιοι και να πληρώνονται από όλους. Αυτό χρειάζεται ισχυρά ευρωπαϊκά στάνταρτ διεξήχθη συζήτηση το προηγούμενο ε, μήνα στο ΕΚΟΦΗΝ και μάλιστα δημόσια συζήτηση. Δεν ξέρω αν μπορέσατε να την παρακολουθήσετε. Θα είχατε δει τότε ποιε είναι οι διάφορε θέσει και τα διάφορα θέματα που απασχολούν του υπουργού. Σα ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι ήταν μια ενδιαφέρουσα ανταλλαγή απόψεων. Τέθηκαν πάρα πολλά θέματα. Έχει μεγάλη σημασία αυτό που είπατε στο τέλος και αυτό που ξεκινήσατε να κάνετε, δηλαδή το πώς θα προχωρήσουμε σε απλούστευση των δημοσιονομικών μας κανόνων. Υπάρχουν δηλώσεις προθέσεων, αλλά προς το παρόν εγώ δεν βλέπω να έχει υπάρξει κάποια ειδική μεταχείριση της Γαλλίας φέτος Ας δούμε λοιπόν πώς ε, εξελίσσονται τα πράγματα βασισμένοι στα δεδομένα, στα γεγονότα. Βλέποντας και κάνοντας λοιπόν, σας ευχαριστούμε για ό,τι κάνατε. Να επαναλάβω και την τελευταία ερώτηση. Νομίζω ότι έχει σημασία η ομοφωνία στο θέμα το φορολογικό. Υπάρχει μια τεράστια προσπάθεια από την Ολλανδική Προεδρία ως προς αυτό το καλωσορίζουμε, το αναγνωρίζουμε. Φυσικά είμαστε περισσότερο φιλόδοξοι και υπάρχουν νέες προκλήσεις για την Ένωση έτσι ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα θέματα της φοροαποφυγής με αποτελεσματικό τρόπο. θα έχουμε συνέχιση νομίζω της καρποφόρου συνεργασίας μας. Okay. Ωραία, σημείο 6 μέρες διάταξη συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την, ε, το πριγκιπάτο του Μονακό για μέτρα ισοδύναμη με αυτά που έχει η οδηγία 2003-48 εισηγητής Αντρέα Σουάμπ Παρακαλώ Ευχαριστώ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι από το Ευρωγκρουπ σε φορολογικέ συμφωνίε που έχουν μεγάλη σχέση και μεγάλη σημασία για τα κράτη-μέλη. Συμφωνία μεταξύ τη Ευρωπαϊκή Ένωση και του Μονακό για κανόνες που περιέχονται στην, ε, στην Οδηγία 48 για την ε, φορολόγηση των τόκων. Όπως ξέρετε και όπως ξέρουν και οι συνάδελφοι, η Ευρωπαϊκή Ένωση έκανε μια συμφωνία για την αυτόματη ανταλλαγή προφοριών για οικονομικά θέματα, για να αποφευθεί η φοροδιαφυγή. Για αυτήν την ιδιαίτερα μικρή χώρα. Είναι η συνέχεια της έκθεσης που είχαμε ήδη εδώ και ε, μερικούς μήνες συζητήσει για το Λίχτενστάιν και άλλες χώρες. Άρα επαναλαμβάνουμε μια, ένα εγχείρημα που ήδη Έχουμε ολοκληρώσει για άλλες χώρες στις 22 ε, Οκτωβρίου μονογράφηκε και ελπίζω να υπογραφεί μόλις φωνεί στο Συμβούλιο. Από τον Ιανουάριο 17 η ενημέρωση για, την, ε, ε, για τις δοσοληψίες που κάνουν οι οι ε, πολίτες της Ένωσης στο Μονακό και αντίστροφα θα είναι υποχρεωτική και θα αρχίσει να... η ανταλλαγή προφορών το 18. Θα ενημερωθούν λοιπόν όλα αυτά. Μέσω της προηγούμενης συμφωνίας είχαμε επιτύχει το Μονακό να δίνει τις ίδιες προφορίες που δίνουμε και εμείς. Η ενημέρωση είναι αναγκαία, διότι η συμφωνία, επειδή έχει αλλάξει το κοινοτικό πλαίσιο το 2014, το TAX 2 λόγω των τελευταίων διεθνών εξελίξεων στον τομέα της αυτόματης ανταλλαγής προφοριών σε επίπεδο ΩΣΑ. Η συμφωνία λοιπόν πρέπει να ενημερωθεί λόγω αυτών των εξελίξεων. Χαιρετίζω αυτή τη συμφωνία όπως και τις άλλες συμφωνίες γιατί μετά τις συμφωνίες με την Ελβετία, την Ανδόρα, το Σαν Μαρίνο και το Λίχτενστάιν είναι άλλο ένα βήμα ούτως ώστε όλα τα κράτη της Ευρώπης να καταπολεμούν την φορολογική απάτη. Με τον ίδιο τρόπο, ενιαία αυτή η ανταλλαγή πληροφοριών για τα στοιχεία των λογαριασμών θα διευκολύνει τις εθνικές αρχές εάν θέλουν πραγματικά να συνεργαστούν, ούτως ώστε να αποφευχθεί η φόρο διαφυγή. Και να είναι και αποτρεπτικά μέτρα ουσιαστικά αυτά, ούτως ώστε να μην κρύβονται ε, περιουσιακά στοιχεία στο εξωτερικό. Στο, προς το συμφέρον μας είναι να επικυρωθεί τάχιστα αυτή η συμφωνία και επειδή θα αξιοποιήσουμε την απλουστευμένη διαδικασία του άρθρου 50 για την έκθεση. Νομίζω ότι η Επιτροπή μας μπορεί να εγκριθεί χωρίς τροπολογίες. Αλλά σας υπενθυμίζω, Πρόεδρε, ότι δεν έχω πρόθεση να αποδεχθώ μέσω της ε, έκθεσης να εισαγάγουμε φράσεις που υπονομεύουν την έκθεση. Και δεν καταλαβαίνω γιατί επετράπει αυτό σε προηγούμενες εκθέσεις. Δεν έχει έννοια οι Ευρωπαίοι νομοθέτε μέσω απλουστευμένη διαδικασία να εγκρίνουν ένα νομοθέτημα αλλά η γνώμη του εισηγητή να περιέχει επιχειρήματα που αντιτίθενται. Δεν έχει καμία έννοια, ούτε διαδικαστική ούτε πολιτική. Γι' αυτό εγώ δεν θα το επιτρέψω. Θα αξιοποιήσω αυτήν την απλουστευμένη διαδικασία ω έχει. Και οι συνάδελφοι που έχουν κάνει αυτέ τι ύποπτε μανούβρες στο παρελθόν ελπίζω να εγκρίνουν την έκθεση μου. Ευχαριστώ πολύ. Thank you. Ευχαριστώ πολύ. Σοσιαλιστική ομάδα, η κυρία Μπερές. Ευχαριστώ. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη από τον σκιώδη μας, τον κύριο Κόφοντ, ο οποίος ψηφίζει στην Επιτροπή Βιομηχανίας. Θέλω να συγχαρώ τον Αλεξάνδρ Σφάμπ για ένα σημαντικό βήμα στη συνεργασία με το Πριγκιπάτο στα πλαίσια της απλουστευμένης διαδικασίας έτσι ώστε να διευρυνθούν οι συμφωνίες που έχουν γίνει με άλλες χώρες όπως το Λίχτενστάιν σε επίπεδο ανταλλαγής πληροφοριών η πορεία που προτείνει ο εισηγητής είναι καλή και η ομάδα μας δεν θα δημιουργήσει πρόβλημα στην ψηφοφορία. Ευχαριστώ πολύ. Λούντς, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και τον εισηγητή. Όπως και προηγουμένως είναι θετική η πρόταση αυτή, θα μας αποτρέψει να αποφύγουμε διπλά μέτρα και σταθμά και θα στηρίξουμε την πρόταση. Σύντομα, να ευχαριστήσω τον Άλεξ για τη δουλειά του. Οι προτάσεις του είναι θετικές. Εγώ η εκλογική μου περιφέρεια είναι στα σύνορα με το Πριγκιπάτο και πρέπει να πάμε σε αυτήν την ωραία περιοχή για να εφαρμόσουμε επιτόπου την εφαρμογή των κανόνων. Δεν έχω κάτι να προσθέσω σε σχέση με αυτό. Έχουν υπάρξει αντίστοιχες εκθέσεις τις οποίες εγκρίναμε. Θετικό εγκρίνουμε. Ευχαριστώ. Μπάρμπαρα. Ο εισηγητής θα ήθελε να πει κάτι να συμπληρώσει. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ναι. Νομίζω ότι λέχθηκαν όλα. Πρόκειται για απλουστευμένη διαδικασία, δεν χρειάζεται και πολύ μεγάλη συζήτηση. Όμω, το βασικό πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε εν προκειμένου είναι το ερώτημα πώ μπορούμε να επιτύχουμε ώστε να, επιτύχουμε μια ε, σε βάθος συνεργασία των εθνικών φορολογικών αρχών. Δεν μπορούμε να τις αναγκάσουμε ούτε και με τις διερευνητικές εργασίες της Επιτροπής για τα έγγραφα του Πάναμα. Το ερώτημα μένει πού μπορούμε να τα βάλουμε τα πράγματα αυτά σε ένα τομέα όπου οι χώρες μέλη έχουν δική τους αποκλειστική αρμοδιότητα. Όχι μόνο λοιπόν να συμφωνήσουν, αλλά και να συνεργαστούν πραγματικά και αποτελεσματικά. Πώ μπορούμε λοιπόν να διαμορφώσουμε τη συνεργασία στο να το επιτύχουμε αυτό. Νομίζω ότι τούτη εδώ η συμφωνία αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προ την κατεύθυνση αυτή και νομίζω ότι η Επιτροπή Οικονομικών πρέπει να εμείνει και να παρακολουθεί διαρκώς πώς λειτουργεί η συνεργασία μεταξύ των εθνικών φορολογικών αρχών. Δεν αναμένω να σημειωθούν σημαντικά προβλήματα σχετικά με την πορεία της εκθέσεως. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος Κουαλτιέρη. Ολοκληρώνεται λοιπόν η συζήτηση εδώ. Σήμερα λοιπόν... Α, ε, για σήμερα τελειώσαμε. Τώρα, η ε, προθεσμία για την υποβολή ενστάσεων έχει παρέλθει. Μπορούμε να θεωρήσουμε λοιπόν ότι εγκρίνεται η έκθεση και να προωθηθεί στην δεύτερη ολομέλεια του Ιουνίου για την τελική ψηφοφορία. Σας ευχαριστώ. Το υπαριθμόν 7 τώρα. Για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και την πράσινη βίβλο. Ο κύριος Λούντβικσον. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σήμερα συνεχίζουμε την εργασία μας για την πράσινη βίβλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις ελληνικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες για ιδιωτικούς πελάτες και μικροκαταθέτες. Αυτό έχει ενδιαφέρον, ε, πράσινη βίβλο δηλαδή έχει ενδιαφέρον, διότι είναι ένας νέος τρόπος αντιμετώπισης νομοθεσίας, πιο δυναμικός και κυρίως θέλουν να συνεργαστούν. Δηλαδή ε, ο στόχος είναι η συνεργασία. Θα συζητήσουμε το σχέδιο της εκθέσεως. Θα κάνω βέβαια και εγώ ό,τι μπορώ για να προχωρήσουν οι συζητήσεις με τους σκιώδεις συζητητές με επικοδομητικό τρόπο. Το σχέδιο εκθέσεως διαιρείται σε τρία τμήματα. Το πρώτο τμήμα περιλαμβάνει γενικές διαπιστώσεις. Το δεύτερο μέρος συζητεί το τι μπορεί και τι πρέπει να γίνει πρόθεσμα. Και στο τρίτο μέρος έρχομαι περισσότερο στο, στις μακροπρόθεσμες προοπτικές. Πρώτα λοιπόν ε, μια διαπίστωση, ότι δηλαδή στην πράξη μένουν ακόμα πολλά να γίνουν για την καταγραφή δεδομένων και ανάλυση τους ενδεχομένως να πρέπει να αυξηθούν οι δυνατότητες που διαθέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επ' αυτού. Και η βάση του, της πράσινης βίβλου δεν είναι αρκετά στέρεα. Χρειαζόμαστε καλύτερη εμπειρική βάση για να μπορούμε να λειτουργήσουμε νομοθετικά με μεγαλύτερη ακρίβεια. Δηλαδή να παραγάγουμε νομοθεσία που να είναι πιο στέρεα. Θα ήθελα επίσης να τονίσω ότι τώρα έχει έρθει η ώρα να λάβουμε συγκεκριμένα μέτρα. Και πρώτα θα πρέπει να απαλληφθεί οποιαδήποτε διακριτική μεταχείριση στην βάση του τόπου διαμονής ή του τόπου κατοικίας. Συχνά οι πελάτες βρίσκονται εντός μιας εθνικής αγοράς και δεν έχουν πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά. Γι' αυτό ο πελάτης θα πρέπει να μπορεί να έχει μπροστά στα μάτια του ολόκληρη την ευρωπαϊκή αγορά. Και σε ό,τι αφορά τον σχεδιασμό της, ε, της ε, προτάσεως θα πρέπει να παραμεριστεί οποιοδήποτε στοιχείο γεωγραφικού αποκλεισμού και να προταθούν εναλλακτικέ δυνατότητες για τον χρηματοπιστωτικό τομέα. Εκτός αυτού θα πρέπει η ευρωπαϊκή αγορά στο σύνολό τη να λειτουργεί με τέτοιον τρόπο ώστε να έχει ο ε, τελικός καταναλωτής ή πελάτης να έχει τη δυνατότητα να συγκρίνει τιμές και προϊόντα. Αλλιώς δεν θα λειτουργήσει ο μηχανισμός αγοράς όπως πρέπει. Στη σύγκριση ποιότητας και τιμών υπάρχουν περιφερειακές ιστοσελίδε που δεν αρκούν όμως γιατί δεν περιλαμβάνουν ολόκληρη την ευρωπαϊκή αγορά. Χρειαζόμαστε λοιπόν μια ε, διαδικτυακή πύλη πανευρωπαϊκή που να επιτρέπει την πρόσβαση σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή αγορά. Είμαι ευέλικτος ό,τι αφορά την δημιουργία αυτή τη δικτυακή πύλη. Αλλά κάτι πρέπει να γίνει. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συντάξει ένα σχέδιο δράσεως. Αλλά τι μορφή θα πρέπει να έχει αυτό. Για παράδειγμα, μπορεί να ληφθεί ως βάση η οδηγία για τις πληρωμές. Τρίτο, οι κανόνες και η πρακτική σε ό,τι αφορά την ταυτοποίηση των όσων ε, στοιχείων θα έχουν ε, σημασία για τη μελλοντική ευρωπαϊκή αγορά πρέπει να γίνει με θετικό τρόπο και να είναι δυνατό να ταυτοποιείται το άτομο και πέραν των συνόρων. Όμως, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι χώρες μέλη πρέπει και στον κανονισμό ΕΝΤΑ να μπορούν να ταυτοποιούνται. Επίσης, να καταβληθεί προσπάθεια ώστε να είναι να ενισχυθεί η ασφάλεια των διαδικασιών για τους ε, καταναλωτές. Τέλος δε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να προβεί σε ανάλυση των συστημάτων αυτών που επιτρέπουν την πληρωμή με πιστοτικές κάρτες σε περίπτωση που υπάρχουν διαφορετικές συναλλαγματικές ισοτιμίες. Εκεί τα πράγματα είναι περίπλοκα και πρέπει να απλοποιηθούν διότι καμιά φορά είναι πραγματικά εξαιρετικά δυσχερές να έχει κανείς ε, εικόνα των διαφόρων συναλλαγματικών ισοτιμιών. Θα πρέπει λοιπόν να προωθήσει μια συνεπή λύση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε ο καταναλωτής να μπορεί να ελέγχει και να κατανοεί την κατάσταση. Πέμπτον, πρέπει κανείς να καταβάλει προσπάθεια για να εξασφαλίσει ώστε και πιο μικρές επιχειρήσεις να μπορούν να έχουν πρόσβαση στην ε, ενιαία αγορά χωρίς εμπόδια. Εδώ μπορούν να υπάρξουν διάφορα μέτρα. Για παράδειγμα, ένα δίκτυο επαφών μεταξύ των χωρών μελών. Ένα, μια μοναδική θηρίδα, ένα one-stop shop. Να μπορούν δηλαδή όσες επιχειρήσεις επιθυμούν να εκμεταλλευτούν τις δυνατότητες που δίνει η ενιαία αγορά, να το επιτύχουν. Αυτά πρέπει να ενταχθούν σε μια ενιαία ατζέντα. Και χαίρομαι που η Πράσινη Βίβλος μπορεί να χρησιμεύσει και ως αφετηρία και για, άλλα, και για άλλες πτυχές. Αναμένω με ενδιαφέρον τις περαιτέρω εργασίες επί του σχεδίου και ελπίζω ότι εν τέλει θα ε, βγει μια ξεκάθαρη και ισχυρή εκθέση που θα υποστηρίξουν οι περισσότεροι δυνατοί βουλευτέ. Ευχαριστώ τον εισηγητή. Κυρία Κούμπνερ, εγώ αντικαθιστώ τον εισηγητή μας τον Σκιώδη, ο οποίος δεν μπορεί να είναι μαζί μας σήμερα. Θα ήθελα ξεκινώντας λέγα ότι η έκθεση αυτή είναι ε, πάρα πολύ καλή έκθεση. Ευχαριστώ τον Λουτβίξον και ε, θα πρέπει να καταφέσουμε μια πολύ φιλόδοξη πρόταση για τις λιανικές οικονομικές υπηρεσίε. Αυτό είναι κάτι το οποίο ανταποκρίνεται με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη δημιουργία της ψηφιακής ενίας αγοράς, όπως επίσης και της Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, Κεφαλαίων είναι θέματα αυτά τα οποία έθεσε ο κ. Λούβιξον που έχουν ε, θα έλεγα καλυφθεί εν πολλής από νομοθετικές προτάσεις τα τελευταία χρόνια και γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι εφαρμόζονται πλήρως οι νομικές αυτές ρυθμίσεις πριν προτείνουμε νέες. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε επίσης να ποσοστοποιήσουμε τα πραγματικά αποτελέσματα και τις επιπτώσεις αυτών των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και γι' αυτό η συλλογή των δεδομένων είναι κυρίαρχη. Η ευρωπαϊκή αγορά στον τομέα των λιανικών αυτών υπηρεσιών είναι ένα μεγάλο κομμάτι των μικρομεσαίων κυρίως και των νέων επιχειρήσεων και επίσης τίθεται το θέμα των επιπτώσεων της ψηφιοποίησης σε πάρα πολλούς τομείς το άνοιγμα των ε, λιανικών αυτών υπηρεσιών σε περισσότερο ανταγωνισμό θα έχει θετικά αποτελέσματα και σε σχέση με τη μείωση των τιμών και σε σχέση με την επιλογή των προϊόντων και σε σχέση με την καινοτομία. Τα εμπόδια στις διαμεθοριακές συνεργασίες στον τομέα αυτών των λιανικών υπηρεσιών είναι σημαντικά. Ακούμε διάφορα εμπόδια σε επίπεδο τυπικό, νομοθετικό, δικαστικό, ε, καθεστώτα προστασίας, ε, δικαστικές αποφάσεις, διαφορετικές συμβάσεις, διαφορετικές γλώσσες. Νομίζω ότι με την ψηφιοποίηση εν μέρη κάτι τέτοιο θα αντιμετωπιστεί και νομίζω ότι υπάρχουν όμως προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν στο μέλλον. Δεν μπορούμε να καλύψουμε τις ανάγκες όλων ε, με τις λιανικές αυτές υπηρεσίες. Υπάρχουν διαφορετικοί τομείς, διαφορετικοί πρωταγωνιστές με τα ειδικά τους χαρακτηριστικά όλοι. Οι μικρομεσαίες ιδιαίτερα αντιμετωπίζουν πολύ υψηλότερα εμπόδια, έχουν συγκεκριμένες ανάγκες και η ευρωπαϊκή αγορά για τις λιανικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες θα πρέπει να επιτρέπουν στις επιχειρήσεις αυτές να έχουν καλύτερη πρόσβαση στην χρηματοδότηση, να διευκολύνονται οι διαμεθοριακές δραστηριοποιήσεις μικρομεσαίων και να υπογραμμίσω εδώ και την ανάγκη να προσφέρουμε στους Ευρωπαίους πολίτες προστασία στον τομέα αυτό, όπως επίσης και την προστασία των προσωπικών τους δεδομένων και των δικαιωμάτων τους σε όλη την Ευρώπη. Γι' αυτό λοιπόν τα κράτη-μέλη πρέπει να εφαρμόσουν τα την οδηγία για τα εθνικά συστήματα προστασίας των καταθέσεων. Μια ευρωπαϊκή αγορά λιανικών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών ε, μπορεί να γίνει με μια αποτελεσματική και αποδοτική νομοθετική ρύθμιση σε εθνικό επίπεδο για την προστασία των δεδομένων. Σχετικά τώρα με τις εγγυήσεις των δικαιωμάτων, το FinNet θα πρέπει να ενημερωθεί και είναι μια ενδιαφέρουσα λύση μην ξεχνάμε ότι η εμπιστοσύνη των καταναλωτών έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και απαραίτητη προϋπόθεση. Η πρόταση των εισηγητών είναι, ε, του εισηγητή μάλλον είναι ενδιαφέρουσα και η εφαρμογή του ΕΝΤΑ, όπως επίσης και οι μονοαπευθυντικές θηρίδες είναι θέματα τα οποία θα πρέπει να τονιστούν στο μέλλον. Θα πρέπει επίσης να δούμε τι γίνεται και σε σχέση με τις επενδύσεις. Οι Ευρωπαίοι πολίτες είναι πιθανοί επενδυτές. Πρέπει να προωθήσουμε την καινοτομία δημιουργώντας κίνητρα για τις επιχειρήσεις να καινοτομούν σε πολλούς τομείς. Επίσης ε, θα πρέπει να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε προϊόντα πανευρωπαϊκού χαρακτήρα. Νομίζω ότι θα συμφωνήσουμε με τις προτάσεις του εισηγητή νομίζω ότι θα μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό σε εύθετο χρόνο. Θα συνεχίσω να συνεργάζομαι και με τους συναδέλφους των υπολείπων πολιτικών ομάδων για να καταλήξουμε σε μια φιλόδοξη πρόταση. Πρέπει να στείλουμε ένα ισχυρό μήνυμα στους καταναλωτές, τους επενδυτές, τις μικρομεσές. Νομίζω ότι η ευρωπαϊκή αγορά στις λιανικές υπηρεσίες, στις χρηματοπιστωτικές πρέπει να οδηγήσει σε μεγαλύτερη εμπιστεσίνη, χαμηλότερο κόστος και καινοτομία. Για να το πετύχουμε αυτό απαιτούνται όμως πολλά νέα βήματα. Ευχαριστώ πολύ. Σάντερ Λούντς για το ίσια ευχαριστώ Πρόεδρε, αντικαθιστώ την ε, Ashley Fox που δυστυχώς δεν μπορεί να παρευρεθεί. θα, τον κύριο Φόξ. Ε, ο κύριος Φόξ υποστηρίζει διάφορα, είναι υπέρ διαφόρων στοιχείων της ε, έκθεσης. Πρέπει να ενισχύσουμε την εσωτερική αγορά για να έχουμε καινοτόμα προϊόντα, περισσότερο ανταγωνισμό και αυτό που είναι ο κύριος στόχος μας, ε, χαμηλότερες τιμές. Συμφωνεί, όπως είπε και η κυρία Χούμπνερ, ότι πρέπει να στηρίξουμε τις καινοτόμες μικρομεσαίες να υποστηρίξουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για να μειώσουν το κόστος τους και άρα να περάσει αυτή η μείωση του κόστους και για τους καταναλωτές. Πιστεύουμε λοιπόν ότι βοηθάνε αυτές οι ρυθμιστικές προσπάθειες για να αναπτυχθούν οι καινοτόμες επιχειρήσεις. Ιδιαίτερα τον ικανοποιεί αυτή η αναφορά σε αυτήν την ενιαία υπηρεσία, one-stop shop. Πολλά γίνονται για αυτό το θέμα. Άρα πρέπει να δούμε πώς θα συντονίσουμε καλύτερα τις προσπάθειες που γίνονται. Υπάρχουν ήδη αυτά τα ενιαία σημεία επαφής ε, στα πλαίσια της οδηγίας για τις υπηρεσίες και μέσω του δικτύου Solvit και λειτουργούν καλά. Άρα δεν θα πρέπει να υπάρξει επικάλυψη. Να έχουμε το πιο αποτελεσματικό σύστημα. Παρ' όλα αυτά, ο κύριος Φόξ έχει και κάποιες ανησυχίες για ορισμένα σημεία της έκθεσης. Πρώτον, έχει αφιβολίες για το ότι το αίτημα για μια ενιαία αγορά για ενυπόθεκα δάνεια είναι περίπλοκος τομέας. Πρέπει να κάνουμε σωστή ανάλυση των επιπτώσεων μιας τέτοιας προσπάθειας, να δούμε τι αλλαγές θα επιφέρει η οδηγία για τα ενυπόθηκα δάνεια πριν υπάρξει περαιτέρω νομοθετική πρωτοβουλία. Να δούμε συνολικά το θέμα και όχι μόνο μία πλευρά. Δεύτερον, λέει η έκθεση ότι πρέπει να υπάρξουν περαιτέρω νομοθετικές πρωτοβουλίες για να σταματήσουν αδικαιολόγητη γεωγραφική αποκλεισμοί. Και αυτό πρέπει να το δούμε με μεγάλη ευαισθησία. Και η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει ότι οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες δεν πρέπει να περιληφθούν στον κανονισμό για τον γεωγραφικό αποκλεισμό. Γιατί οι γεωγραφικοί παράγοντες ε, είναι στοιχεία του προφίλ κινδύνου του καταναλωτή. Άρα πρέπει να υπάρξει διαβούλευση και με τα κράτη-μέλη. Για τις ορισμένες περιπτώσεις ε, η άρνηση παροχής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών μπορεί να είναι ιτολογημένη. Σε άλλες όχι γιατί κάποιοι εμπορικοί παράγοντες πρέπει, ε, συγγνώμη, μπορεί να επηρεάσουν το κόστος ε, κάποιας υπηρεσίας και η κατάσταση είναι διαφορετική μεταξύ διαφόρων δικαιοδοσιών, άρα πρέπει να το δούμε αναπερίπτωση. Τρίτον, τρίτο σημείο ανησυχίας. Αυτή η ιστότοπη ε, συγκρίσεων ίσως είναι λίγο νωρίς. Αν δεν έχουμε περισσότερα προϊόντα που να μπορούν να απολυθούν ε, διαμεθοριακά, ε, δεν ξέρω τι έννοια έχει να ευαισθητοποιήσουμε περισσότερο τους καταναλωτές. Αλλά αυτό είναι περισσότερο θέμα χρονικής στιγμής. Και, εν πάση περιπτώσει, ο κύριος Φόξ προσλέπει στην περαιτέρω συνεργασία με τους κοιόδης και τον εισηγητή για την βελτίωση του κειμένου. Ευχαριστώ πολύ. Ο Πρόεδρος. Και εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω και εγώ. Θα... Δεν θα μιλήσω Ολλανδικά αντικαθιστώντας τη Σόφιντ Τίντφελτ, αλλά θα συνεχίσω στα αγγλικά. Νομίζω ότι μια ενιαία αγορά στις λιανικές υπηρεσίες τις χρηματοπιστωτικές έχει τεράστιες προοπτικές. Πρέπει να είμαστε φιλόδοξοι, πρέπει να είμαστε ταχείς Νομίζω ότι αν χάσουμε το χρόνο μας και διστάσουμε θα χάσουμε τις ευκαιρίες. Πρέπει να προσαρμοστούμε στις αλλαγές, δεν πρέπει να υπάρχουν ταμπού. Τα κράτη-μέλη θεωρητικά και μόνο στηρίζουν τις ενιαίες αγορές, αλλά είναι εθνικιστές πρωταγωνιστές των συμφερόντων των δικών τους πιστοτικών ιδρυμάτων. Νομίζω ότι η ορθολογική νομοθεσία και η σωστή φορολογική αντιμετώπιση των λιανικών προϊόντων των χρηματοπιστωτικών είναι πολλές φορές εμπόδια στις διαμεθοριακές συναλλαγές. Είναι θέμα αυτό το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί, ακόμα και αν γνωρίζουμε ότι τα κράτη-μέλη θα προβάλλουν αντίσταση. Είναι μια αναπόδραστη συζήτηση εφόσον θέλουμε να προχωρήσουμε και θα καταθέσουμε τροπολογίες στην έκθεση. Για το χρονοδιάγραμμα φοβάμαι ότι το χρονοδιάγραμμα δεν θα μας επιτρέψει να βοηθήσουμε ιδιαίτερα το πρόγραμμα δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η έκθεση προς διαβούλευση θα παρουσιαστεί στο τέλος Ιουνίου, το πρόγραμμα δράσης προβλεπόταν το Σεπτέμβριο, αλλά έχει πάει μάλλον το Νοέμβριο. Νομίζω ότι θα πρέπει το ταχύτερο δυνατόν να προχωρήσουμε έτσι ώστε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει υπόψη της απόψεις του Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ. Thank you. Uh, Ευχαριστώ. Ο κύριος Βιέχας για την ΓΟΕ. Ευχαριστώ. Εγώ ε, εκπροσωπώ την ε, σκιώδη συγγήτριά μας, Μαρίζα Ματίας. Έχουν τεθεί ορισμένε ερωτήσει. εδώ συζητήθηκαν με ορισμένα θέματα. Πρώτα, το ερώτημα αν θα πετύχουμε μεγαλύτερη χρηματοπιστωτική ενοποίηση. Όμως όσο μεγαλύτερη γίνεται αυτή, τόσο περισσότερο συγκεντρωτικό γίνεται το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Έχουμε λοιπόν εμείς την ανησυχία ότι μπορεί αυτό να οδηγήσει στην δημιουργία μεγάλων χρηματοπιστωτικών ολιγοπολίων. Κάτι που θα είναι σε βάρος τελικώς και των καταναλωτών και των πολιτών. Αυτό είναι ένα δίδαγμα το οποίο θα έπρεπε να είχαμε διδαχθεί από την κρίση. Μετά έχουμε και ορισμένα αιτήματα. Η πράσινη βίβλος προσπαθεί να συγκεράσει διάφορες απόψεις, τα συμφέροντα του χρηματοπιστικού συστήματος με τα συμφέροντα του τελικού καταναλωτή. Αλλά δεν νομίζω να είναι αυτός ο σωστός δρόμος. Οι τράπεζες έχουν το καθήκον να δημιουργούν χρηματοπιστωτικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Όμω πρώτο το καθήκον του είναι η προστασία των καταναλωτών. Εξάλλου, σημειώνεται και σημαντική πίεση στους ε, τραπεζικούς υπαλλήλους που βρίσκονται στην άμεση επαφή με τον πελάτη. Το ερώτημα είναι εάν θα δίνονται οικονομικά κίνητρα στους ε, ανθρώπους αυτούς αλλά αυτό δεν είναι θεμελιώδε. Θεμελιώδε είναι να γίνει η παρέμβασή μα στη συνολική στρατηγική των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Φαίνεται να υπάρχει και η ψευδέστηση εδώ μεταξύ ορισμένων ότι ο μεμονωμένος καταναλωτή που συνήθω δεν γνωρίζει τι πραγματικότητε των χρηματοπιστωτικών συστημάτων εάν στη διάθεσή του περισσότερε πληροφορίε θα είναι η στέση να κατανοήσει καλύτερα την αγορά ότι θα είναι δηλαδή διαφανέστερη η αγορά. Όμως, αν θέλουν πραγματικά, αν θέλουν πραγματικά ρεαλιστικά να προστατεύσουμε τον καταναλωτή, πρέπει τότε να διαγραφούν ορισμένα προϊόντα και να μην πολλούνται, διότι είναι πολύ περίπλοκα και προκαλούν δράματα χρηματοπιστωτικά προϊόντα τα οποία έχουν καταστρέψει οι οικογένειες τους, έχουν στερήσει και τις τελευταίες αποταμιεύσεις τους, δράματα τα οποία τα έχουμε δει στην Πορτογαλία. Η Πράσινη Βίβλος αναγνωρίζει ότι οι καταναλωτές νιώθουν βαθιά δυσπιστία απέναντι στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Και μετά μιλούν για όλο και μεγαλύτερη συγκέντρωση, που κατά τη γνώμη μας δεν είναι ο σωστός δρόμος. διότι ανοίγει το δρόμο, αυτός ο δρόμος, αν μπορώ να το πω έτσι, σε όλο και μεγαλύτερες καταχρήσεις από τα ολιγοπόλια. Ευχαριστώ. Γκίγκουλτ. Ευχαριστώ. Και ευχαριστώ και τον Όλο Λούτζικσον για την καλή έκθεσή του. Νομίζω ότι είναι θαυμάσια βάση για να τοποθετεί το Κοινοβούλιο και φυσικά συμφωνώ με αυτά που είπαν η Σοφή και η Σιλβή ότι πρέπει να τοποθετηθούμε έγκαιρα για να ακουστεί η φωνή μας επί της ουσίας βεβαίως ισχύει ότι οι επενδυτές λαμβάνουν ένα πολύ μικρό τμήμα ε, από τα κέρδη που προκαλούνται από τις ε, χρηματοπιστωτικές ε, ενέργειες και ένα πολύ μεγάλο τμήμα πηγαίνει στους ενδιάμεσους. Οπότε, βεβαίως πρέπει να υπάρξει περισσότερος ανταγωνισμός, ούτω ώστε το κόστος της διαμεσολάβησης θα μειωθεί. Βεβαίως, σωστό μου φαίνεται. Αλλά κοιτάξτε, πρέπει να είμαστε και ειλικρινεί μεταξύ μα. Τι σημαίνει να υπάρξει ανταγωνισμό για να μειωθεί το κόστο των ε, ενδιαμέσων. Και δεν νομίζω ότι είναι απόλυτα ειλικρινή η Κομισιόν με τον τρόπο με τον οποίο να αντιμετωπίζει το θέμα. Διότι. Γιατί οι καταναλωτέ δεν εμπιστεύονται κάποια προϊόντα τα οποία εκδίδονται σε άλλε αγορέ, Εδώ συμφωνώ απόλυτα με το ΕΛΚ. Υπάρχουν τεράστιες διαφορές όσον αφορά τη φορολόγηση, τον πτωχευτικό νόμο, τις νομικές προϋποθέσεις. Δεν ε, εμπιστεύεσαι κατά ανάγκη έναν ενδιάμεσο σε άλλη χώρα. Άρα οι νομικές βάσεις θα πρέπει τουλάχιστον να εναρμονιστούν σε τέτοιο βαθμό που να δημιουργηθεί κλίμα εμπιστοσύνη. αυτό είναι το πρώτο. Άρα πρέπει να δούμε ακριβώς το πλαίσιο. Συμφωνώ με τον εισηγητή είναι θέμα εάν ως καταναλωτής θεωρείς ότι θα αντιμετωπιστείς σωστά. <clears throat> και πρέπει λοιπόν να υπάρχει το ίδιο επίπεδο προστασίας του καταναλωτή σε όλες τις χώρες για να έχει εμπιστοσύνη σε κάποιο προϊόν που εκδίδεται και πωλείται αλλού. Δεύτερον, αν τα προϊόντα διαφέρουν σε κάποιες μικρές λεπτομέρειες, δεν είναι εύκολο να τα συγκρίνεις και ούτε θα βοηθήσουν οι στότοποι σύγκριση. Πρέπει να είναι παρόμοια τα προϊόντα. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει περισσότερη τυποποίηση των προϊόντων. Για παράδειγμα, τα συνταξιδοτικά προϊόντα. Αλλά αν θέλουμε να υπάρξει ανταγωνισμός, όπως και σε άλλου κλάδους που υπάρχουν υψηλά περιθώρια κέρδους, χρειαζόμαστε ευρωπαϊκού ορισμού των βασικών στοιχείων κάθε τέτοιου προϊόντος, των βασικών χαρακτηριστικών. Επίσης, αν κάποια προϊόντα είναι ε, συνδεδεμένα με το ένα με το άλλο, είναι δύσκολο να τα συγκρίνουμε. Πρέπει λοιπόν ως κοινοβούλιο να είμαστε, ως κοινοβούλιο, να είμαστε ε, απόλυτα ειλικρινείς και να μην εκφράζουμε απλώς κάποιες επιθυμίες. Πρέπει να πούμε ποιες πρέπει να είναι οι βασικές προδιαγραφές σε όλους αυτούς τους τομείς. Αν θέλουμε πραγματικό διαμεθοριακό ανταγωνισμό για να μειωθούν τα περιθώρια κέρδους των ενδιαμέσων. Για να μειωθούν οι διαστάσεις αυτού του συστήματος ενδιαμέσων που είναι τερατώδης. Διότι αν δεν υπάρχει ανταγωνισμός για αυτό το κόστος της διαμεσολάβησης, βραχυπρόθεσμα προστατεύουμε κάποιες ε, υπηρεσίες ενδιαμέσων, αλλά τελικά το FinTech θα το κάνει πιο αποτελεσματικά και δεν θα εδρεύει στην Ευρώπη αλλά αλλού. Υπάρχει λοιπόν προστατευτισμός για αυτές τις ε, ε, υπηρεσίες διαμεσολάβησης που είναι παραφουσκωμένες. Πρέπει να κάνουμε λοιπόν μια ειλικρινή συζήτηση για την επιτήρηση της προστασίας των καταναλωτών στα χρηματοπιστωτικά πλήματα, γιατί έχουμε το ίσας. E αλλά το ίσας e δεν έχει πόρους για να επιτηρεί, για να επιβλέπει. Ενώ στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχει ένα, μια υπηρεσία με ίδιους πόρους για την επιτήρηση της προστασίας των καταναλωτών. Δεν θα υπάρξει εμπιστοσύνη στα διαμεθοριακά προϊόντα εάν δεν υπάρχει εμπιστοσύνη στην επίβλεψη της προστασίας του καταναλωτή. Και κάτι άλλο που είναι πολύ σημαντικό είναι τα πράσινα χρηματοπιστωτικά προϊόντα είναι σημαντικά για τους καταναλωτές. Όπως και στο PRIPS με την Περβάνς και την ΣΥΡΠΑ είναι θα πρέπει ακριβώς να δημιουργήσουμε κοινούς κανόνες για το πρασίνισμα των προϊόντων σε αυτόν τον κλάδο και ελπίζω και ο Σουηδός συναδελφός μου να ε, ε, βλέπει θετικά το πρασίνισμα του κλάδου αυτού της οικονομίας και πιστεύω πραγματικά το έχω εμπιστοσύνη ότι θα έχει. Δεν βλέπω τον Μάρκο Βάλλη με το Catch the Ευχαριστώ. Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω τον Όλε για την πρότασή του. Είναι μια πολύ καλή βάση συζήτησης πάνω σε ένα θέμα στο οποίο λόγω των πρωτοβουλειών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν έχουμε προχωρήσει παρά μόνο πάρα πολύ επιφυλακτικά με ελάχιστες νομοθετικές παρεμβάσεις. Τέσσερα σημεία. Κατανοώ ότι η γενική αντιμετώπιση από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι μια προσπάθεια διευκόλυνσης ε, των λιανικών υπηρεσιών. Κανένας δεν μπορεί να είναι εναντίον, εφόσον είναι προς όφελος των ε, καταναλωτών. Υπάρχουν όμως κάποιες εγγυήσει εδώ, οι οποίες θα έλεγα είναι απαραίτητες. Έχοντας υπόψη είναι αυτά τα οποία έχουμε κάνει σε σχέση με το ΚΡΙΠΣ. Νομίζω ότι θα συμφωνήσω με τον εισηγητή. Θα επιδιώξουμε να υπάρξει μια συγκρισιμότητα ανάμεσα στα διαφορετικά προϊόντα. Μία από τις προτάσεις τις οποίες κάνω, όταν βλέπουμε αυτά τα οποία κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση ε, με την οδηγία για τα δελτία, νομίζω ότι θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε σε ένα τυποποιημένο δελτίο, σαν γι' αυτό που είπαμε στα κρύψη, για να διευκολύνουμε τη συγκρισιμότητα. Αυτοί που ασχολούνται με τα δελτία πολλές φορές μας λέγουν ότι η περίληψη αυτή νομίζω ανήκει σε μια διαφορετική λογική, είναι κάτι το εντελώς διαφορετικό. Εγώ νομίζω ότι ένα τέτοιο δελτίο είναι κάτι το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο για τους επενδυτές σε λιανικές υπηρεσίες. Η δεύτερη παρατήρηση την οποία θα ήθελα να κάνω είναι ότι η Ευρωπαϊκή στο παρελθόν είχε κάνει μια πρόταση για την δυνατότητα ενός μηχανισμού αποζημίωσης των επενδυτών. Το κοινοβούλιο μας υπό την ευθύνη του συναδέλφου Σμιτ είχε εκφραστεί υπέρ μια τέτοιας Ρύθμιση. το Συμβούλιο όμως δεν θέλησε να το συζητήσει αυτό και από τότε το θέμα βρίσκεται σε στασιμότητα. Αν θέλουμε όμως να ξανακερδίσουμε την εμπιστοσύνη των πελατών για τις λιανικές υπηρεσίες, πρέπει να υπάρξει ένας μηχανισμός αποζημίωσης σε περιπτώσεις λάθους, σε περιπτώσεις κακών συμβουλών από τους ε, λειτουργούντες στην αγορά. Τρίτη παρατήρηση είναι το θέμα της διανομής των προϊόντων αυτών μέσω διαδικτύου. Πολλοί συνάδελφοι ε, έθεσαν το θέμα του FinTech. Έχουμε πράγματι σήμερα κάποια προϊόντα τα οποία διανέμονται από το διαδίκτυο που οδηγούν σε καταχρήσει εις βάρος των καταναλωτών απαράδεκτες. Είμαι βεβαία λοιπόν ότι είναι ευθύνη της Επιτροπής να κάνει πιο συγκεκριμένες προτάσεις. Και τέλος, σε σχέση με την εποπτεία της προστασίας των καταναλωτών, ε, τα στοιχεία είναι στη διάθεση των υπηρεσιών των εποπτικών, Παρ' όλα αυτά περιμένουμε πάντα την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε πολλούς τομείς. Εμείς προχωρήσαμε σε σχέση με τα PRIPS. Εδώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να συμπληρώσει με νέες προτάσεις τις οποίες περιμένουμε γιατί αποτελούν τμήμα του συνόλου των προτάσεων που θα μας επιτρέψουν να προχωρήσουμε θετικά. Ευχαριστώ πολύ. Δεν υπάρχουν άλλοι ομιλητές. Συνεπώς ξαναδίνω το λόγο στον Όλε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα πρώτα να ευχαριστήσω τις και τους συναδέλφους για τις παρεμβάσεις. Βεβαίως ένα πράγμα είναι σίγουρο, υπάρχουν κάποια εμπόδια τα οποία πρέπει να εξαλειφθούν. Και όπως είπα υπάρχει η βραχυπρόθεσμη και η μακροπρόθεσμη πορεία με τον στόχο να φροντίσουμε ώστε να μπορεί να λειτουργήσει το σύστημα διαμεθοριακά. Άρα να ενισχυθεί και ο ανταγωνισμός. Και αυτό θα οδηγήσει εν τέλει στο να μπει στο επίκεντρο ο καταναλωτής. Για δε μικρές και μεσές επιχειρήσεις είναι σημαντικό να έχουν στη διάθεσή τους μια διαμεθοριακή αγορά. Αυτά θα χρειαστούν χρόνο, χωρίς αμφιβολία. Θα προσπαθήσω να προχωρήσω όσο γίνεται πιο όσο γίνεται με ταχύτερο ρυθμό για να μπορέσουμε να καταθέσουμε την κοινή μας πρόταση έγκαιρα για να μπορέσουμε να επηρεάσουμε τα όσα θα προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ λοιπόν για όλες τις προτάσεις. Ευχαριστώ και εκ των προτέρων για τις τροπολογίες που θα καταθέσετε και τις οποίες βέβαια θα επεξεργαστώ και θα κάνω κάθε το δυνατόν ώστε να επιτύχω μια ευρεία πλειοψηφία σε επί εγγράφου που να καταθέσουμε εδώ στην Επιτροπή και μετά να αποχωρήσει και στην Ολομέλεια. Ελπίζω και είμαι και βέβαιος ότι όλα θα πάνε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ο πρόεδρος Γκουαλτιέρη. Το χρονοδιάγραμμα έχει ω εξή Κατάθεση τροπολογιών έως τις 28 έκτου το μεσημέρι. Εξέταση τροπολογιών μέχρι 31 Αυγούστου ψήφος στην ΕΚΟΝ 29 Σεπτεμβρίου και στην Ολομέλεια, στην πρώτη Ολομέλεια του Νοεμβρίου. Ευχαριστώ πολύ. Εδώ ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του σημερινού πρωινού και ξαναρχίζουμε στις 3 με τον Επίτροπο κύριο Χίλ.